Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θέλω να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων ε, της Σλοβενίας, τον κύριο Μπόμπερ, για να μας μιλήσει για τις εργασίες του Διεθνούς Ταμείου Αρρωγής για την εκαθάριση ναρκοπαιδείων και την παροχή βοήθεια σε θέματα ναρκών. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που συχνά πυκνά το αναφέρουμε και στην Επιτροπή μας και το οποίο έχει ιδιαίτερη έτσι, απήχηση σε, ένα, σε μια περιοχή που η όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια που και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία problème de nature technique. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μάλλον με τη διερμηνία τι γίνεται. Parfait francophone. No. Βέβαια, ξέρετε όλοι από ό,τι κατάλαβα τέλεια γαλλικά, έτσι. Qu'est-ce qui se passe Ah, le Slovène est sur le canal anglais. C'est une évolution intéressante. oui, oui c'est bon Ok. Bien. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Το διεθνές λοιπόν αυτό ταμείο ε, για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Μπαγκαρίμπα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ε, κυρίως πολύ σημαντική περιοχή για την κοινή πολιτική για την ΚΕΠΑ και Γίνονται και αρκετές αποστολές εκεί, Κωσυφοπαίδιο, Βοσνία Ζεγοβίνη, έχουν σημαντικές προσπάθειες γίνει. Ο κύριος Μπόκα, λοιπόν, υπουργό Εξωτερικών, ζήτησε και από τον συνάδελφο Πάσκο, αντιπρόεδρο, να συμπροεδρεύσει. Φυσικά και θα εστιάσουμε στις ε, δράσεις ναρκοθέτησης, αλλά θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το πεδίο μας. Ο κύριος Μπάγκαρ, από ό,τι ξέρω, θα μπορούσε να εντάξει αυτή την ε, πρωτοβουλία και στο πλαίσιο της ευρύτερης ε, πολιτικής ε, της Σλοβενίας στην περιοχή αυτή. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε την εισαγωγική παρέμβαση του Υπουργού και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση. Θα ζητήσω όμως πρώτα από τον κύριο Πάσκου να μας κάνει μία εισαγωγή. Θέλω απλά να καλωσορίσω τον Υπουργό και να πω ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλιά του. Λοιπόν, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο θέμα με τη μετάφραση. Ε, μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό. Lep pozdrav eh, eh, Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας μιλήσω Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μου δίνεται η δυνατότητα να σας μιλήσω για το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής ε, για την απομάκρυνση ναρκών. Αυτό το Ταμείο Αρρωγής συστήθηκε από κοινού με τη Σλοβενία και τις άλλες χώρες περιοχής. Και το Ταμείο αυτό ασχολείται με θέματα απομάκρυνσης ναρκών. Στη δική μου λοιπόν την ομιλία θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσω να σας ε, εξηγήσω ε, την εξωτερική πολιτική της ε, Σλοβενίας και πώς ακριβώς αυτό το Ταμείο Αρρωγής προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Ε, βέβαια, τα θέματα βρίσκονται εν εξελίξη και ε, το Ταμείο Ρογής, το ITF όπως το λέμε εν συντομία, είναι ένα πρόγραμμα που πλέον έχει καταξιωθεί. Ε, το Ταμείο αυτό Ρογής ε, δεν ασχολείται με όλα τα θέματα της πολιτικής, κατ' ουσίαν ασχολείται με τα βασικά θέματα της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής της Σλοβενίας. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τρεις βασικές έννοιες, τρεις στόχους αν θέλετε, που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της Σλοβενίας. Και κατόπιν θα εξηγήσω, θα προχωρήσω πώς ακριβώς εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο οι δραστηριότητες του Ταμείου Αραγής. Οι βασικές αρχές είναι ε, η ηθική, η παγκοσμιότητα και τρίτος στόχος είναι να υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια. Θα σας εξηγήσω σύντομα πώς ακριβώς ε, αντιμετωπίζουμε αυτούς τους τρεις βασικούς στόχους. Καταρχήν, όσον αφοράμε για μια ηθική εξωτερική πολιτική, εμείς προσπαθούμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος ε, στο διεθνές σκηνικό, ακολουθώντας και αρχές όπως είναι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη ε, και ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές που καθορίζουν τις θέσεις μας στην εξωτερική πολιτική. Ας δούμε τώρα λιγάκι ε, πού εντάσσεται ε, το θέμα του Ταμείου Ραγής. Ε, οι νάρκες ξηράς και οι μη εκραγέντες εκρηκτικοί μηχανισμοί του πολέμου έχουν βεβαίως μακρόχρονα αποτελέσματα για τους πολίτες γιατί εξακολουθούν να παρακολύουν την επιστροφή των προσφύγων, την ανοικοδόμηση, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση των χωρών που πλήττονται από αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει η σύμβαση της ΟΤΑΒΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει σημαντικά στην απομάκρυνση αυτών των αρκών για να παρεμποδίσει και τι προεκτάσει του σε ανθρώπινο επίπεδο. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει περισσότερο από όλου του άλλου ε, στην εξουδετερώση των αρκών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, Προσπαθούμε να συνεχίσουμε την ανοικοδόμηση, το Ταμείο Αρρωγή για την Απομάκρυνση Ναρκών. Όπω είπαμε, η συντομία ITF συστήθηκε το Μάρτιο του 1988 από την κυβέρνηση τη Σλοβενία πριν κάνει στη Σλοβενία επικυρώσει τη συνθήκη τη Οτάβα. Εν τω μεταξύ, το Ταμείο Αρρωγή επεξέτεινε τι δραστηριότητέ του ε, από τη Σλοβενία, επεκτάθηκε σε όλε τι χώρε τη περιοχή. Χώρε που πλήττονται από το πρόβλημα των ναρκών. Όλε αυτέ την περιοχή πλήττονται και επεξέτεινε τι δραστηριότητε του και πέρα από ε, την ε, στενή έννοια της περιοχής. Θα μου επιτρέψετε τώρα να επανέλθω στην ε, ηθική πολιτική, εξωτερική πολιτική όπως την ανέφερα, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας ηθικής εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκα και στη θέση που έχουμε λάβει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα ψηφίσματα και τις θέσεις που εκφράσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ανθρωπίνων Εθνών, όπου ήμασταν μέχρι πρόσφατα μέλος. Οι θέσεις μας αυτές αφορούν κυρίως τη Μέση Ανατολή. Ε, εξάλλου, οι θέσεις μας αφορούν ε, και ε, τα γεγονότα στην Γάζα και στην Φρουτίλια όπως επίσης ε, και όλες τις άλλες ε, θέσεις ε, που έχουμε εκφράσει σχετικά με το Παλαιστινιακό. Η εξωτερική μας πολιτική περιλαμβάνει και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ισχυρότερη παρουσία κυρίως στην Παλαιστίνη και κυρίως φέτος, όπου βλέπουμε πλέον να έχουμε φτάσει στην τελική φάση του Παλαιστινιακού. Όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική, συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμεθα σε όλους τους τομείς προστασίας ανθρωπινών δικαιωμάτων, κυρίως όσον αφορά την προστασία ευάλωτων ατόμων, γυναικών και παιδιών που εμπλέκονται σε διενέξεις και αργότερα θα σας εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες ε, το πρόγραμμα της Γάζα, το οποίο έχει επιληφθεί το Ταμείο αλλά θα ήθελα να φέρω και δραστηριότητες που ε, συνεχίζουμε για την κατάσταση στο Νταφούρ, όπου ε, πριν από αρκετά χρόνια ο πρώην Πρωθυπουργό μας είχε ασχοληθεί με την κατάσταση στο Νταφούρ και με την κατάσταση των πολιτών στην περιοχή αυτή, στον Ταφούρ. Άλλα θέματα που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου είχαν σχέση με την ε, περιφερειακή αλλά και την ε, παγκόσμια διάσταση της ε, εξωτερικής μας πολιτικής. Όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής μας, ε, εδώ αναφέρομαι στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σλοβενία εξακολουθεί να είναι ένθερμος οπαδός ε, της ε, ένταξης όλων των χωρών της περιοχής στο ΝΑΤΟ. Για το στόχο αυτό εμείς συμβάλλουμε πολιτικά, οικονομικά αλλά και στρατιωτικά και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό μη φιδόμενοι κόπου και προσπαθειών. Υπάρχει η συμφωνία ανάμεσα στη Σλοβενία και την Κροατία για τα σύνορα, μια συμφωνία που ετέχθη σε ισχύ την προηγούμενη χρονιά. Η συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ μόλις η ε, Σλοβενία υπογράψει τη Συμφωνία Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της περιφερειακής συνεργασίας. Ε, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία για αυτό το θέμα της διευθέτησης των συνόρων και κάνοντας αυτό το βήμα ενισχύσαμε τη συνεργασία με την Κροατία. Ε, συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμεθα σε σημαντικά πολιτικά φόρουμ στα Δυτικά Βαλκάνια, ε, σε διάφορες ε, αποστολές από τη Γιούλεξ μέχρι την UPM και την Αλτέα. Και βεβαίως συμμετέχουμε και στην K4 όπου έχουμε διαθέσει ε, ένα σημαντικό τμήμα ανδρών της Σλοβενίας. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία απελευθέρωσης της χορήγησης θεώρησης, ε, χαιρόμαστε που ολοκληρώθηκε πέρυσι η διαδικασία. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα της κατάργησης θεώρησης ε, και θεωρούμε ότι ε, πρέπει οι πολίτες ε, να μπορούν να μετακινούν ελεύθερα στην Ευρώπη, ακριβώς όπως συνέβαινε πριν από 20 χρόνια. Η εμπειρία μας από την κατάργηση της θεώρησης κατέδειξε πόσο σημαντική ήταν αυτή η κίνηση για τους νέους κυρίως, αλλά και γενικότερα για τους πολίτες περιοχής. Οι νέοι βεβαίως αποτελούν το μέλλον. Η ευρωπαϊκή προοπτική παραμένει το σημαντικότερο κίνητρο ε, για τις χώρες περιοχής για να ε, εξελιχθούν περαιτέρω, για να προβούν σε μετερρυθμίσεις και θέλω να πω ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι η κινητήρια δύναμη των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια όπως συνέβη και με τη δική μου τη χώρα όταν εμείς ε, θελήσαμε πριν από κάποια χρόνια να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστη ε, προοπτική στις χώρες αυτές. Βεβαίως και οι ίδιες οι χώρες οφείλουν και εκείνες ε, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά εφέτος, χρειαζόμαστε μια ημερήσια διάταξη. Τι θέλει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή ε, για την χρονιά του 2011. Υπάρχουν διάφορες φάσεις που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αφήσουμε κατά μέρο την Κροατία, για την οποία ελπίζουμε ότι ε, θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις και θα υπογραφεί εφέτος η συνθήκη ένταξης, κατά τα άλλα έχουμε χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο επίπεδο πάντα κάτω από το πρίσμα της ενταξιακής διαδικασίας. Ε, μπορούν αυτές βέβαια ε, να ενταχθούν σε κάποιες ομάδες, χωρίς αυτό είναι επίσημο. Έχουμε μία ομάδα κρατών οι οποίες προχωρούν. Ε, έχουμε τη Μακεδονία η οποία ε, περιμένει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Έχουμε το Μαυροβούνι που είναι υποψήφια χώρα και επίσης ελπίζουμε ή ελπίζει η χώρα ε, μέχρι το τέλος να πάρει μια ημερομηνία και έχουμε και τη Σερβία η οποία πρόκειται σύντομα να καταθέσει το ερωτηματολόγιο και θεωρούμε ότι και αυτή θα προχωρήσει με ταχύτητα ε, στην ε, ενταξιακή διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν ε, χώρες ε, για τις οποίες ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές ε, διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η μία ομάδα και κατόπιν υπάρχει και μία άλλη ομάδα όπου έχουμε την Αλβανία η οποία κατέθεσε αίτηση ένταξης και η οποία περιμένει να χαρακτηριστεί υποψήφια χώρα. Κατόπιν έχουμε την Βοσνία Ερσεγοβίνη που ακόμα δεν έχει καταθέσει αίτηση ένταξης και έχουμε και το κοσφοπέδιο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει αναπτύξει σχέσεις ούτε έχει παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα κρατών ε, για τα οποία ελπίζουμε ότι και αυτά θα προχωρήσουν. Ελπίζουμε ότι ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Εμείς ε, ως ε, Σλοβενία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ο Πρωθυπουργό μας έχει ορίσει ειδικό εντεταλμένο για τη Βοσνία για να μπορέσουμε και να τους ε, κατανοήσουμε καλύτερα και να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Γιατί θα ήταν τραγικό για μια χώρα που υπέφερε περισσότερο από όλους τους άλλους από τον πόλεμο να ε, παραμείνει καθυστερημένη πιο πίσω στην ενταξιακή διαδικασία όπως συμβαίνει τώρα. Εφόσον μιλώ για τα Δυτικά Βαλκάνια, θα ήθελα να σας μιλήσω πού ακριβώς εντάσσεται το Ταμείο Αρρωγής για την εξουδετέρωση ναρκών. Όπως σας εξήγησα προηγουμένως, ε, το Ταμείο Αρρωγής ξεκίνησε ως Ταμείο Αλλαγής καταρχήν για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κατόπιν όμως επεξέτεινε τις ε, δραστηριότητες του στην ευρύτερη περιοχή και ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξετέρωση απομάκρυνση ναρκών ε, στην Μακεδονία, στο Μαυροβούνι, ε, στη Σερβία και υπάρχουν δύο χώρες όπου εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τις ενάρκειες. Οι χώρες αυτές είναι η Βοσνία, και η Κροατία. τα περισσότερα κονδύλια τα οποία συγκέντρωσε κατά τα τελευταία έτη το ε, Διεθνές Ταμείο Αρρωγής για την Εκαθάριση Ναρκοπαιδείων, τα χρήματα αυτά ε, διοχετεύτηκαν στις περισσότερο πληγήσεις χώρες. 150 εκατομμύρια ευρώ έχουν ε, δοθεί από το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής για την Εκαθάριση Ναρκοπαιδείων στην Βοσνία και ένα εξίσου σημαντικό ποσό διατέθηκε για τον ίδιο σκοπό στην Κροατία το Διεθνέ Ταμείο Ρογή έχει δρομολογήσει και την περιφερειακή συνεργασία στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη για την εκαθάριση ναρκοπεδίων. Οι δραστηριότητε του, οι δραστηριότητε που αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή, στηρίχθηκαν από το Διεθνέ Ταμείο Ρογή και αυτό κρίθηκε σε ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, ανάμεσα στι χώρε που ε, ξέφυγαν από τι διενέξει. Ουσιαστικά αυτή είναι και η πρώτη επαφή των χωρών αυτών. Το πρώτο θέμα επί το οποίο συνεργάστηκαν μετά τον πόλεμο ήταν δηλαδή το θέμα της εκαθάρισης ναρκοπαιδίων. Και ε, κατόπιν ε, προέκυψε ένα είδος ε, συμβουλίου, συντονιστικού συμβουλίου Αργότερα το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής ήταν κέντρο ε, αριστείας ε, για την εκαθάριση ναρκωπεδίων Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ε, στηρίζουν την περαιτέρω δραστηριοποίηση του Διεθνούς Ταμείου Αρρωγής και πέρα από την στενή έννοια της περιοχής. Το Διεθνές Ταμείο εμπλέκεται σε παρεμφερή προγράμματα στη Μέση Ανατολή, στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία. Το 2009 ο ΣΑ και το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής ε, δρομολόγησαν από κοινού ένα πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα της εκαθάρισης ναρκοπαιδίων με στόχο τις διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες χώρες στην Κεντρική Ασία και με το Αφγανιστάν για να υπάρχει περιφερειακή συνεργασία παραμπερίς με αυτή που ε, προέκυψε στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα υπάρχει λοιπόν ένα Συμβούλιο Συντονισμού Εκαθάρισης Ναρκοπαιδίων στην Κεντρική Ασία. Ε, αυτή θα είναι και η συνεργασία ανάμεσα στο δικό μας, το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής για τα Βαλκάνια και το, το Συντονιστικό Συμβούλιο που θα προκύψει για την Κεντρική Ασία. Πάντα με στόχο την εκαθάριση ναρκοπαιδίων. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να συνεχίσω με το τρίτο θέμα με, τις, ε, με τη τρίτη δέσμη αρχών που καθορίζουν την ε, εξωτερική πολιτική της Σλοβενίας, η οποία είναι φιλόδοξη, Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι πολίτες. Καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την ε, ζωή των ανθρώπων, ε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για σταθερότητα και ευμάρεια. Το Ταμείο Αρρωγής, το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής, συστήθηκε ως ένα πρόγραμμα το οποίο θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, και αργότερα ε, θα ήθελα να σας αναφέρω και συγκεκριμένα στοιχεία πόσα τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή εκαθαρίστηκαν και επίσης ε, θα σας ε, αναφέρω και στοιχεία ε, πέρα από τη δική μας περιοχή. Το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής συντονίζει και το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Γάζα. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την αποκατάσταση παιδιών θυμάτων στη Γάζα. Μέχρι τώρα λοιπόν το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής έχει βοηθήσει στην αποκατάσταση 51 παιδιών από τη Γάζα, 9 ψυχασθενείς, εκείνο λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν στη Λουμπιάννα, εκείνο το οποίο πράττει το Διεθνές Ταμείο Ρογής είναι το ότι φέρνει τα παιδιά από τη Γάζα και αυτό το πράττει σε συνεργασία με ε, Παλαιστινίους επιτόπου, τοπικούς φορείς. Φέρνουμε λοιπόν τα περισσότερο πληγέντα παιδιά, τα οποία έχουν χάσει ε, ένα ή δύο μέλη τα φέρνουμε στη Σλοβενία για αποκατάσταση. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε 120 παιδιά από τη Γάζα. Τα παιδιά αυτά ε, μένουν στη Σλοβενία τρεις με τέσσερι εβδομάδες και κατόπιν επιστρέφουν στη Γάζα. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση της πρωτοβουλίας μας. Ε, δηλαδή, ε, το Διεθνέ Ταμείο Ρογή συνεργάζεται με τις παλαιστινιακέ Αρχές για να ε, οικοδομηθεί ένα κέντρο αποκατάστασης επιτόπου στην ίδια την Παλαιστίνη και εκεί να συνεχίζεται η αποκατάσταση των θυμάτων ε, το Παλαιστινιακό Κέντρο Αποκατάστασης κάποια στιγμή μάλιστα να αναλαμβάνει πλήρως την αποκατάστασή τους χωρίς να χρειάζεται τα παιδιά αυτά να έρχονται στη Σλοβενία. Σε μια μεταγενέστερη φάση ενδιαφερόμεθα να οικοδομήσουμε σχολεία. με την ΟΝΡΑ, η οποία συμμετέχει επίσης σε προγράμματα στη Γάζα. Κατά κάποιον τρόπο, αν θέλετε δηλαδή, προσφέρουμε ολοκληρωμένη ε, ψυχοσωματική αποκατάσταση και κοινωνική αποκατάσταση των παιδιών. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα ε, το οποίο μπορεί να είναι μικρής κλίμακας, όμως ε, ένα πρόγραμμα που επιφέρει κολοσιαίες αλλαγές στα παιδιά θύματα. Μιλώντας για την ε, φιλόδοξη και ουσιαστική εξωτερική πολιτική που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να αναφέρω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανακτήσουμε την ε, μη μόνιμη θέση μας ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα έτη 12 και 13. Αυτή είναι μια πραγματική επιθυμία της Σλοβενίας. Η Σλοβενία επιθυμεί να κάνει χρήση της εμπειρίας της, ε, της εφαρμογής προγραμμάτων, των γνώσεών της, γιατί προσπαθούμε ε, να δώσουμε απαντήσεις σε κοινά ε, προβλήματα ή αν θέλετε κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ε, κάποια στοιχεία που αφορούν ε, στο Διεθνές Ταμείο Αρρωγής για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα τι ακριβώς κάνει το Ταμείο αυτό. Από τότε που προέκυψε είχαμε πάνω από 130 δωρητές οι οποίοι συνέβαλαν ε, στους πόρους του Διεθνούς Ταμείου. 28 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της UNDP. Το ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο το οποίο συγκεντρώνει πόρους από διάφορους, ε, διάφορα μέρη. Πρόκειται για ένα επιτυχημένο διατλαντικό πρόγραμμα για τη λειτουργή με δωρεές ε, των Ηνωμένων Εθνών που συνδυάζονται με δωρεές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο και όλα αυτό, το σύνολο του ποσού διοχετεύτηκε για την εκαθάριση ναρκοπαιδίων. Το 1998 ξεκινήσαμε ως ένα μικρό ταμείο αρρωγής, αλλά λόγω του χαμηλού διοικητικού κόστους του ταμείου και λόγω του ότι οι δωρητές ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του ταμείου, το ταμείο εν συνεχεία ανέλαβε όλες τις δραστηριότητες εκαθάρισης ναρκοπαιδίων στα Δυτικά Βαλκάνια. ...107 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στα Δυτικά Βαλκάνια εκαθαρίστηκαν ε, με τη βοήθεια του Διεθνούς Ταμείου... ...και 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στον Νότιο Κάφκασο. Περισσότεροι από χίλιοι ε, συμμετείχαν στις δραστηριότητες ε, και ενημερώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών ε, για την καθάριση των αρκοπαιδίων. Τώρα το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής εφαρμόζει μια νέα στρατηγική η στρατηγική αυτή εκτείνεται από το 2009 μέχρι το 2013. Μιλάμε για δραστηριότητες ακαθάρισης, αλλά και παροχής βοήθειας στα θύματα κάτω από το πρίσμα της ανθρώπινης ασφάλειας. Ε, προσπαθούμε να στηρίξουμε και τις ε, συμβάσεις καταστροφήν όπλων και πυρομαχικών παράλληλα με δραστηριότητες που αναπτύσσουμε στον τομέα της ασφάλειας, ε, στον αφοπλισμό ε, και στην επανένταξη. Αυτοί είναι οι τομείς ε, στους οποίους αναπτύσσουμε δραστηριότητες. Θα ολοκληρώσω λοιπόν την παρέμβασή μου και θέλω να πω ότι οι νάρκες ξηράς είναι υπολείμματα περασμένων παλαιών εποχών και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καταστροφή τους. Θα ήθελα να εκφράσω τις, ε, την, τις μου προς την αμέριστη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολλών ευρωπαϊκών κρατών, βοήθεια που προσφέρουν τα κράτη αυτά ε, στο Διεθνές Ταμείο Αρρωγής. Ε, συνεχίζουν να προσφέρονται κονδύλια στο Ταμείο για να συνεχίσει και αυτό να αναπτύσσει τις δραστηριότητε του καθάριστα ναρκοπαιδείων στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και σε άλλες περιοχές. Ε, για όλους αυτούς του λόγους το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής θεωρούμε ότι είναι ένα επιτυχημένο πείραμα που αποδείχθηκε στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση έχω τέσσερα αιτήματα. Θα ήθελα να σας εκτιμήσω ότι το 2011 είναι μια σημαντική χρονιά για τη χώρα σας. Τον Ιούνιο γιορτάζεται την 20η επέτειο της ανεξαρτησίας σας. Έχουμε δύο Σλοβαίνους βουλευτές μεταξύ μου από σήμερα που δραστηριοποιούνται ε, ο κύριος Βάγγελ που συνεισέφερε τα μάλα και ο κύριος Κάτσιν που είναι και για την Σερβία. Αναφερθήκατε επίσης στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για κατάρριση θεωρήσεων ε, διαβατηρίου. Η κυρία Τάνια Φάγιν είναι υπεύθυνη εδώ και έχει εργαστεί πολύ στο Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Πέτρελε βέβαια έχει κάνει πολλά, δεν είναι, απόψε, δεν είναι σήμερα συγγνώμη, μαζί μας, αλλά έχει κάνει και αυτός ε, πάρα πολλά και στο πλαίσιο της πολιτικής μας και την κεντρική Ασία. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Σλοβαίνοι βουλευτές είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος μιας χώρας. Μπορούν πολύ καλά και μικρές χώρες να κάνουν πολύ ποιοτική δουλειά. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανόρντεν, ο οποίος είναι υπεύθυνο εισηγητής για το Mine Action. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Λοβενίας και να τον ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος για τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ στις δράσεις ε, για την Σνάρκες. Ε, όπως είπε και ο πρόεδρος, είμαι εισηγητής για ένα έγγραφο, ένα ψήφισμα αν θέλετε, για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε ό,τι αφορά τη δράση στον τομέα των ναρκών ε, ε, τα προηγούμενα χρόνια. και για το ITF ήμουν τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκανα και εγώ πολλά για να συγκροτηθεί αυτό το ταμείο. Η δράση στον τομέα των ναρκών είναι ένα από του τομεί νομίζω ότι που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει καλή δουλειά. Όπως είπατε και εσείς ε, είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης. Το Ταμείο Ρογή ε, ήταν κάτι πολύ θετικό, γιατί υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα στα Βαλκάνια που έπρεπε να αντιμετωπιστεί και εσεί φαίνεται ότι έχετε μια καλή προσέγγιση, ιδίω και με την ε, συγκέντρωση πόρων από τι ΗΠΑ και χαίρομαστε ιδιαίτερα με την επιτυχία σας και θέλουμε να σας συγχαρούμε για το έργο το οποίο επιτελείται εδώ και αρκετά χρόνια. Πρέπει να πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπω όπως και οι διεθνεί οργανισμοί, ε, όταν εγκατασταθούν κάπου δεν φεύγουν ποτέ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και αυτούς τους οργανισμούς όταν μιλάμε για τις δράσεις μας στον τομέα ε, των ναρκών. Γνωρίζετε την Ανατολική Ευρώπη <clears throat> και την ε, Βοσνία Ζεγοβίνη και ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας ε, σε ποιο βαθμό υπάρχει ακόμη πρόβλημα ναρκών και θυμάτων από νάρκες σε αυτό το μέρος του κόσμου. Όταν συμφωνήθηκε το 1997 η συνθήκη της Αχρίδας, ε, κάποιοι δεν είχαν ε, δια πιστό ή συνειδητοποιήσετε πρόκειτο για μια διεινική διαδικασία. Είχαμε κάποιες ιδέες στο μυαλό μα ε, για μια δεκαετία. Νομίζαμε ότι είναι ένα επαρκέ χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στους τομεί προτεραιότητας για την ε, βοήθεια των, ε, στα θύματα από νάρκες και στην καθάριση του ναρκοπεδίου. Αν δει κανεί αυτή την περιοχή, τη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τόσο έντονη παρουσία και δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόσα πολλά πράγματα να γίνονται, να έχουν γίνει. Εσείς είπατε ότι το πρόβλημα σχεδόν έχει περκεραστεί. Πάντοτε όμως ε, θεωρούσα ότι δεν έχουμε παρκώς χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών οι οποίες ήταν σε εμπόλεμη σύραξη και μιλώ συγκεκριμένα για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, όπου φαίνεται να υπάρχει απροθυμία να συμμετάσχουν ενόπλε δυνάμεις, αλλά ξέρετε στι περιοχέ αυτέ μιλάμε για αυτού που είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι για την ναρκοθέτηση. Αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν και την ε, μείζωνα ευθύνη και υποχρέωση από ναρκοθέτηση, σε καθάριση των ναρκοπαιδίων. Φαίνεται να έχουν απροθυμία όμω να το πράξουν. Και νομίζω ότι έχουμε χάσει μια ευκαιρία Θέλω να σας ρωτήσω αν ε, είναι και σε ποιο βαθμό είναι αποδέκτης κοινοτικών κονδυλίων ακόμη το Ταμείο Αρρωγής και πώς ε, ε, στηρίζεται αυτό το ταμείο. Θα με ενδιαφέραν βέβαια και πολλά άλλα από αυτά που κάνετε. Είπατε ότι έχετε επεκτείνει τις δραστηριότητές σας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο επίκεντρο για μας η περιοχή αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε λύσαμε το πρόβλημα, κλείσαμε και τα μαζεύουμε. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που πρέπει να γίνουν, πάντως σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε και για το καλό έργο που έχετε επιτελέσει και για την παρουσία σας εδώ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Βανόρτεν. Έχουμε τέσσερις ομιλητές, ε, έχουμε στη θέσή μας μέχρι τις 11 και 4. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι λοιπόν για να μπορέσει και ο κύριος Υπουργός να απαντήσει Συνεχίζοντας τα ερώτημα του κύριου Βανόρντεν, θέλω και εγώ να σας ρωτήσω το εξής. Φυσικά στη Βόσνια, Ζεγοβίνη, η ένταση, το εύρος, η εμβέλεια της ε, σύγκρουσης ε, εξηγεί το γιατί δεν έχει ακόμη ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης ναρκοπαιδείων. Τα προβλήματα όμως που έχετε αντιμετωπίσει είναι αμυγός ποσοτικά λόγω της εμβέλειας του μεγάλου αριθμού ή έκτασης των ναρκοπαιδείων ή υπάρχουν και πολιτικές δυσκολίες όπως αυτές που βλέπουμε στη Βοσνία οι οποίες εξηγούν τις καθυστερήσεις που βλέπουμε. Το γεγονός ότι είμαστε ακόμη μακριά από την επίτευξη του στόχου της αποναρκοθέτησης. Κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κύριε Υπουργέ ότι πολύ σωστά αναφερθήκατε ε, στην, ε, στο Ταμείο Αρρωγής ε, ITF ως μια επιτυχία της Σλοβενίας. Όντως και ορθώς επίσης θέσατε το ζήτημα αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζετε και ορθώς το πράτετε τα ναρκοπέδια και τις νάρκες σαν ένα υπόλοιμα πολιτικής του παρελθόντος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, διαφορετικά είδη ναρκών τώρα. Ε, έχουμε ανθρώπους ε, που γίνονται οι ίδιοι νάρκες. Έχουμε αύξηση των τρομοκρατικών ενεργειών και οι ίδιοι οι άνθρωποι γίνονται πλέον νάρκες. Είναι ένα άλλο είδος πολέμου, ίσως πιο τρομακτικό και από αυτές ε, τις ε, κλασικές νάρκες που αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα ήδη. Όσον αφορά την αξιολόγηση του προβλήματος ε, των ναρκών, κυρίως εκεί που στις περιοχές που ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κρίσεις σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να υποψιαστούμε ότι θα υπάρξει αύξηση των ε, ναρκών νέου τύπου, ότι θα υπάρξει αύξηση ε, των κρυφών ενεργειών που με κάποιο τρόπο θα πρέπει να απελευθερωθούν. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γιατί είστε νεότερος πολιτικός ε, και έχετε και την ε, ευθύνη κατά κάποιο τρόπο για την ε, μελλοντική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί προλαλήσατε, έθεσαν κάποια από τα ερωτήματα που είχα σκοπό εγώ να θέσω. Και να προσθέσω και εγώ τότε ένα ερώτημα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ βέβαια τον Υπουργό για την παρουσία του και για τις πολύ ικανοποιητικές εξηγήσει που μας έδωσε. Υπάρχει μια πτυχή που είναι σημαντική σε κάθε πολιτική, ιδίω σε δημοκρατική πολιτική, πολυμερή πολιτική. Η κοινή γνώμη, ο κόσμος, ο λαός. Και νομίζω ότι δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το πρόγραμμα, ε, αυτό του Ταμείου Αρρωγής μεταξύ της κοινή γνώμης και, ε, και εγώ και προσπαθώ και στην Ισπανία να αλλάξω κάποια πράγματα γιατί ε, στις συζητήσει που γινόνται είτε στα πανεπιστήμια είτε σε διάφορα κέντρα έχει ανακύψει το ζήτημα των αρκών Σε μια συγκεκριμένη λοιπόν συζήτηση όταν εγώ αναφέρθηκα στο πρόγραμμα αυτό και στην επιτυχία που έχει ε, κάποιοι έδειξαν κάποιο σκεπτικισμό και συγκεκριμένα και κάποιες πιο ριζοσπαστικές μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις λένε ότι κάποιες χώρες ουσιαστικά κάπως κοροϊδεύουν. Δηλαδή, αντί να δίνουν ε, τους πόρους για την αποναρκοθέτηση, ή ενώ δίνουν πόρους για την αποναρκοθέτηση, συγχρόνως κατασκευάζουν και νέε άρκες, νάρκες. Άρα, ε, πρώτο θέμα, επικοινωνία με την κοινή γνώμη, ενημέρωση της κοινή γνώμη. Δεύτερον, πολύ καλά ε, μας και αγραφήσατε την ε, εικόνα, το πανόραμα της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και τι δυνατότητες υπάρχουν για προσέγγιση, σύνδεση και ίσως και προσχώρηση. Ίσως να μην διαβάζουμε ούτε να ακούμε ούτε να βλέπουμε κάθε μέρα αρνητικές πτυχές ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν θετικές πτυχές που προβάλλονται και έχουμε και έναν ε, κατάλογο μελών που θέλουν να μπουν. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι που θέλουν να προσχωρήσουν, δεν είμαστε πια και μια λέσχη τόσο κακή. Και πιστεύω ότι και η προσχώρηση των μελών θα μας εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λούνατσεκ, η οποία είναι και η συγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Προθέσεων για το Κωσυφοπαίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για ε, την αναφορά που κάνατε στο έργο του Ταμείου Αρρωγής και συγχαρητήρια για αυτά τα οποία έχετε επιτύχει όχι μόνο στη Βοσνία αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλκανικής τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι πολύ σημαντική η δράση σας, γιατί όπως και εσείς ε, ο ίδιος είπατε, η καταστροφή των ε, ναρκοπαιδείων, η αποναρκοθέτηση ε, έχει και κοινωνικές και άλλες διαστάσεις και επιπτώσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μπορεί κανείς να ελαφρύνει τον πόνο αμάχων, ε, τον πόνο απλών πολιτών που υπέφεραν από όλη αυτή την πολεμική διαδικασία. Επίσης ε, η προσπάθεια διασύνδεσης αυτών των προγραμμάτων εκαθάρισης ναρκών από ναρκοθέτησης με αναπτυξιακά προγράμματα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα εκτιμούμε ιδιαίτερα. Μία ερώτηση όσον αφορά αυτές τις νάρκες κατά προσωπικού, τις cluster Minds της ενάρκης διασποράς. Ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο όσον αφορά και την επίτευξη των αρχών της συνθήκης του ε, Δουβλίνου. Εσείς αναφέρεστε, ε, ε, συμπεριλαμβάνετε στην προσπάθειά σας και της νάρκες διασποράς. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γιάννης μόλις πριν, οι δραστηριότητες ε, του ε, Ταμείου θα σας οδηγήσουν και στο να προσπαθήσετε να συζητήσετε με χώρες οι οποίες έχουν απόθεμα ε, βομβών, ναρκών διασποράς, ναρκών καταπροσωπικού, έτσι ώστε να καταστρέψουν το απόθεμα αυτό. Ξέρω ότι πολλά αναφέρονται στη συνθήκη, αλλά κάποιες χώρες δεν ακολουθούν και, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι πόσο πιέζεις αυτές τις χώρες να κινηθούν προς μια κατεύθυνση. Και μια άλλη ερώτηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2006 είχαμε μια έκτακτη γραμμή του προϋπολογισμού για τα ναρκοπαίδια. Αυτό ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Και τα χρήματα πλέον που αναφέρονται στην εκαθάριση ναρκοπαιδείων ε, έχουν πάει σε άλλα κεφάλαια τι προτείνετε εσείς, τι μας συστήνετε να κάνουμε. Να έχουμε μια, ε, μια επιπλέον γραμμή προπολογισμού για τις νάρκες ή να, να, συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα, δηλαδή στο μηχανισμό σταθερότητας να βάζουμε και τα χρήματα για τις ε, νάρκες. Ε, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα μέρος τα χρήματα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα αποκατάστασης και είπατε ότι για το κοσφοπέδιο ε, και είπατε ότι ολοκληρώθηκε το ζήτημα για το κοσφοπέδιο. Ναι, αλλά εγώ λέω, σαν εισηγήτρια και για το θέμα, ε, ότι αποκλείονται οι πολίτες του κοσφοπεδίου. Τέλος, ο κύριος ε, Κατσίνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη Σερβία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως και η συνάδελφος Ουλρίκε μόλις προείπε, υπάρχει ανάγκη να παράσχουμε βοήθεια στις χώρες ώστε να μπορέσουν να αποσταρμολογήσουν τεράστια αποθέματα βαρέων ε, πυρομαχικών που είναι παντού στον κόσμο και όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια. Όταν ήμουν και εγώ μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρρωγής, συζητούσαμε για το πώς μπορούμε να βρούμε κάποια καθοδήγηση και πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις ε, προσπάθειες του Ταμείου πριν έχουμε την έκρηξη του, στην Αλβανία της αποθήκης με τις τρομερές επιπτώσεις που έχει αυτό για τον τοπικό πληθυσμό. Πάντως υπάρχουν αρκετές τέτοιες αποθήκες στην Ευρώπη, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Υπάρχει κάποια σκέψη για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή πολλαπλασιασμού διάδοσης ε, των ε, δραστηριοτήτων ε, του Διεθνούς Ταμείου Αρρωγής προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή είμαστε η υποεπιτροπή για την ασφάλεια και την άμυνα, Ουσιαστικά το θέμα είναι η ασφάλεια και το κλίμα, η ατμόσφαιρα σε μια περιοχή. Είχαμε κάποιες πρόσφατες ταραχές στα Τύρανα και επειδή θρηνήθηκαν ε, θύματα τώρα έχουν κάπως παγώσει τα πράγματα αλλά υπάρχει φόβος ότι μπορούν να επαναληφθούν ε, ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα επεισόδια. Θέλω να ακούσω την άποψη της κυβέρνησής σας πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ λεπτή αυτή η κατάσταση στην Αλβάνια. Φυσικά υπάρχει απελευθέρωση ε, ε, των ταξιδιών με την κατάρρευση θεωρήσεων διαβατηρίου αν όμως είχε συμβεί αυτό το γεγονός πριν από τρεις μήνες, δεν θα υπήρχε καν αυτή η των θεωρήσεων, η απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατήριου. Υπάρχει αυτή λοιπόν η κατάσταση στην Αλβανία. Και σε σχέση με αυτό θέλω να αναφέρω και τη συζήτηση που γίνεται στο Στρασβούργο, την ώρα που μιλάμε, την έκθεση ΜΑΤ, για την διακίνηση οργάνων. Είναι ένα πάρα πολύ επίμαχο έγγραφο, δεν έχει εγκριθεί ακόμη και δηλητηριάζει πραγματικά την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν τεράστιες κατηγορίες και καταγγελίες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διέξοδος, να βρεθεί διέξοδος από τον ε, επικίνδυνο κύκλο, από αυτή τη δίνη που επιταχύνεται. Και όλα αυτά δεν είναι επικίνδυνα μόνο για την Αλβανία και το Κωσυφοπέδιο, αλλά δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και στο Βελιγράδι και επισκιάζουν τις θετικές εξελίξεις στην όλη περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την θέση της δικής σας κυβέρνησης σε σχέση με το εν λόγω έγγραφο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάφτιν ζήτησε το λόγο σύντομα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ και συγχαρητήρια για την ε, εξαιρετική και σημαντική δράση σας σε διεθνές επίπεδο. Έχω μια τεχνική φύσεως ερώτηση, ερώτηση αποσαφήνισης. Κατάλαβα ότι τα χρήματα ξεκινούν και από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες και μετά, δηλαδή μέσα από διάφορους χορηγούς, δωρητές και μετά έχουμε και τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος όμως συντονίζει τις ε, δραστηριότητες, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλο ένα ερώτημα. Στο ITF ε, ασχολείστε και με, τον, ε, με την αγορά του εξοπλισμού ή μονάχα ασχολείστε με το θέμα της αποναρκοθέτησης και της αποκατάστασης ε, των ε, θυμάτων. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες εξοπλισμού, Μποζένα είναι η μία, αν δεν κάνω λάθος, σε Πρόκειται για βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό. Ε, εσείς ασχολείστε και με την αγορά αυτού του εξοπλισμού. Έχετε δικό σας εξοπλισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για την απάντηση. Σας ευχαριστώ για τα θετικά λόγια σας τα, υπέρ, τα λόγια σας υπέρ της δουλειά του Ταμείου. Και πρέπει να σας πω ότι και εμείς στη Σλοβενία είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες μας και με αυτό το Διεθνές Ταμείο Αρρωγής δείχνουμε ότι είμαστε μια μικρή σε διαστάσεις χώρα, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε και να κάνουμε πράγματα που έχουν σημασία και να συνεισφέρουμε σε συγκεκριμένα σχέδια. Να περάσω στα αγγλικά και να αναφερθώ στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ζητώ συγγνώμη γιατί για το κοσυφοπέδιο όντως χρησιμοποίησα λάθος ε, έκφραση. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο κοσυφοπέδιο, μια και μιλάμε για τα Δυτικά Βαλκάνια και το κοσυφοπέδιο είναι ακόμα μέσα. και βεβαίως θα θέλαμε να ε, ξεκινήσει ο διάλογος με το Κωσυφοπέδιο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και είναι σαφές βεβαίως ότι και το Κωσυφοπέδιο εντάσσεται στα Δυτικά Βαλκάνια και ε, επομένως ε, θα πρέπει να ξεκινήσει και ο διάλογος για την θεώρηση εγγράφων, ταξιδιωτικών εγγράφων για τη Βίζα και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και το διάλογο που ξεκίνησε μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, ε, ε, θα πρέπει να ενταχθεί το θέμα αυτό και στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, όσον αφορά την Βοσνία. Το πρόβλημα των ναρκοπαιδίων ε, στην Βοσνία ισχύει ακόμα, το ίδιο και στην Κροατία. Υφίσταται πρόβλημα ναρκών στις χώρες αυτές. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα στάδια Ε, στάδια στην αποναρκοθέτηση και το, ο στόχος μας ε, θεωρητικός είναι το στάδιο 3 των ε, ναρκών. Αυτό είναι το ιδεώδες. Δηλαδή είναι το χωρίς καθόλου νάρκες, αλλά και το mine safe, το στάδιο δηλαδή στο οποίο υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά τις νάρκες, είναι και αυτό ένα ικανοποιητικό στάδιο. Οι περισσότερες χώρες είναι ήδη στο στάδιο mine safe ή mine free. Πάντως, στις χώρες που αναφέραμε προηγουμένως, Βοσνία και Κροατία, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις νάρκες. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία από ναρκοθέτηση στη Βοσνία. Εστιάζουμε την προσοχή μας στα Δυτικά Βαλκάνια και δεν θέλω να σας δοθεί εντύπωση ότι ε, παραμελούμε τα Δυτικά Βαλκάνια για να δραστηριοποιηθούμε σε άλλες ε, περιφέρειες. Απλώς ε, η Σλοβενία και το Ταμείο κοιτάει και προς το μέλλον και βλέπουμε ότι η ανάγκη αποναρκοθέτησης μειώνεται στα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα χρειαζόμαστε και λιγότερα χρήματα για την αποναρκοθέτηση στα Δυτικά Βαλκάνια και επομένως πρέπει να δούμε πού αλλού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λειτουργικό ταμείο ε, για διαδικασίες επαναρκοθέτησης ή ακόμα και για κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την αποναρκοθέτηση. Ε, και σαν επόμενο βήμα θα μπορούσαμε να δούμε τα ελαφρά όπλα, αλλά ε, αυτό όντω είναι ένα επόμενο βήμα. Το Ταμείο Αρρωγής, το ITF, έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση ε, στην χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο ε, εγκαθίδρυσε αφενός η Σλοβενική κυβέρνηση και μετά η κυβέρνηση της Βοσνίας. Επομένως δεν είναι απολύτως επιλέξιμο ε, για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα θα πρέπει ε, να τροποποιηθεί κάπως αυτό το ταμείο έτσι ώστε να δέχεται περισσότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η χρηματοδότησή του μάλλον, ε, λειτουργεί ως εξής το Αμερικανικό Κογκρέσο κάθε χρόνο ε, δίνει κάποια χρήματα για το ITF, για την αποναρκωθέτηση δηλαδή. Και εκεί προστίθενται και χρήματα, από την Ευρωπαϊκή, και χρήματα ευρωπαϊκά. Και μέσω ενός ειδικού προϋπολογισμού ε, τον ε, προϋπολογισμό των Ηνωμένων, Εθνών, με τον, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τον τρόπο αυτό ε, πιο εύκολα μπορούμε να συνδυάσουμε ε, τα χρήματα αυτά με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Τώρα, η όλη κατάσταση στην Βοσνία, ναι, βεβαίως μας ενδιαφέρει. Είχαμε πρώτα απ' όλα τέσσερα χρόνια που χάθηκαν στην ουσία ε, λόγω της προηγούμενης ε, ε, κυβέρνησης. Η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί ως έχει. Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Βοσνία, κάτι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την προσέγγιση μας. Δεν αναφέρομαι στην αποναρκωθέτηση. Αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται κανονικά αλλά εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την Βοσνία. και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε τις τρεις εθνότητες να συνυπάρχουν. Um, Ο κόσμος έχει υποφέρει πάρα πολύ στους, ε, στη διάρκεια των ε, ε, πολέμων, αλλά θα πρέπει πλέον να στρέψουμε την πλάτη μας προς το παρελθόν, σε ό,τι έγινε στη διάρκεια των πολέμων και είναι καλό και για αυτούς, θα είναι καλό και για μας. Αλλά βεβαίως είναι ένα ζήτημα προς σκέψη για όλους μας. Η ερώτηση όσον αφορά τα προβλήματα που δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καιροί και κάποια από τα προβλήματα τα οποία μας δημιούργησαν προβλήματα στο παρελθόν ή μας άφησαν αδιάφορους στο παρελθόν, ε, να πούμε ότι πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση, έχουμε γυρίσει σελίδες. Όλα τα προβλήματα μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν κάτι συμβεί στην ε, Αλβανία, που έχει ήδη κατά κάποιο τρόπο ξεκινήσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας αφορά και μας ενδιαφέρει άμεσα. Στην, ε, για την Αλβανία τι να κάνουμε λοιπόν. Είχαμε μια άτυπη διάσκεψη το Σαββατοκύριακο μεταξύ Υπουργών για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην Αλβανία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να βλέπουμε μονάχα απλώ σαν παρατηρητές την κατάσταση ε, η οποία εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια δράση στην, ε, ε, στην Αλβανία, να έρθουμε σε επαφή με τα πολιτικά κόμματα. Τον Μάιο ε, θα οργανωθούν εκλογές. Θα πρέπει και εμείς να συζητήσουμε με τους εταίρους, να τους βοηθήσουμε, να συζητήσουμε με τα κόμματα που θα προετοιμάσουν τις εκλογές αυτές. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς. Ενδεχομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με, τον, με τους δύο ηγέτες, δηλαδή τον υπεύθυνο της κυβέρνησης και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Ξέρω ότι πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε κάποιες προσπάθειες. Ενδεχομένως πρέπει να ξαναρχίσουμε τις προσπάθειες και πλέον ως Συμβούλιο, ως ε, ε, ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθουμε σε επαφή με τους δύο ηγέτες, να τους ενθαρρύνουμε να συζητήσουν ε, μαζί μας να φωτίσουμε περισσότερο την κατάσταση. Έχουμε ένα νέο πρέσβη στα Τύρανα από πλευράς ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικών ε, Δράσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ορατός αυτός ο πρέσβης, να αναμειχθεί όσο γίνεται περισσότερο. Επανερχόμενο όμως στα προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί, δεν είναι μόνο η Αλβανία φυσικά, στην Μεσόγειο βλέπουμε ότι έχουμε και εκεί εξελίξεις. Μας απασχολεί όλους τα, το, τι γίνεται στην Τίνιδα, στην Τινησία, αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση, αναρωτιόμαστε, μα πώς δεν προβλέψαμε, πώς δεν το είδαμε να έρχεται. Ίσως γιατί δεν υπάρχει αρκετός, ε, αρκετά αναπτυγμένος διάλογος ανάμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τις ε, χώρες αυτές. Και ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε, να ενισχύσουμε το διάλογο το, με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν βρεθεί όμοιροι ε, ε, ε, στην, επίλυση του Παλαιστινιακού. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο ή μπορεί ακόμα καλύτερα να αποτρέψει τέτοιου είδης κρίσεις. Γιατί, ξέρετε, στο τέλος θα είναι δικό μας το πρόβλημα ε, ε, όσον αφορά δηλαδή την, ε, την επίπτωση που θα έχει στη μετανάστευση, στην ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Άρα θεωρώ, εκλαμβάνω την ερώτησή σας σαν ενθάρρυνση στην προσπάθεια επίλυσης όλων των ανοιχτών προβλημάτων από το Κυπριακό μέχρι το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. σχετικά με τις ε, νάρκες ε, διασποράς ε, και την καταστροφή του αποθέματος. Για την ώρα το ITF ασχολείται με τα ναρκοπαίδια και τον καθαρισμό ναρκοπαιδίων και σιγά σιγά αρχίζει να ασχολείται και με τα ελαφρά όπλα. Η προσέγγιση είναι διαφορετική βέβαια όσον αφορά την καταστροφή των ε, ναρκών και την καταστροφή των ε, ελαφρών ε, όπλων. Ας πούμε στην Σερβία γίνεται μεγάλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει ήδη για την απομάκρυνση μη εκραγέντων μηχανισμών ή βομβών. προσπαθούν να αναπτύξουν και την πραγματογνωμοσύνη τους ε, και τις τεχνικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν. Ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει επιπλέον η Σλοβενία έτσι ώστε ή το Ταμείο έτσι ώστε να ε, ενισχυθεί η καταστροφή των αποθεμάτων. Κάνουμε ε, διάφορες, προσεγγίζουμε το θέμα. We are, um, uh, we presented the Το 2012 θα κληθούμε να προεδρεύσουμε τις ε, συνάντηση ε, της διαδικασίας της ΟΤΑΒΑ και στα πλαίσια αυτής της προεδρίας θα σκεφτούμε τρόπους ε, για ε, περαιτέρω απονορκοθέτηση και καταστροφή των αποθεμάτων. Βεβαίως ε, τα Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένας από τους, μία από τις μεγάλες χώρες που ελπίζουμε ότι ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μαζί τους διμερείς συζητήσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μεγάλες χώρες. πρέπει να πούμε ότι έχουμε εξελίξεις ε, και ε, το Κογκρέσο και η ίδια η Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ε, υπέρ της διαδικασίας περαιτέρω συζήτησης. Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ νομίζω ότι μία γραμμή του προϋπολογισμού σαφέστερα θα μπορεί να δείξει πόσα χρήματα υπάρχουν και τι ε, μπορεί να γίνει. Ενώ εάν έχουμε πολλές ε, γραμμές, ε, τότε μπορεί να υπάρχει έτσι και μια κρυφή ατζέντα κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση για την αποναρκοθέτηση μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ότι μειώνεται το ίδιο το πρόβλημα των ναρκών. Άποψή μου λοιπόν θα ήταν να κρατήσουμε μία έξτρα γραμμή του προϋπολογισμού. Ε, τέλος για την έκθεση Μάρτη. Οι καταγγελίες οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρές και έχουν σημαντική επίπτωση επιτόπου. Ε, ελπίζουμε ότι ότι η εργασία αυτή, η έκθεση αυτή αποτελεί ε, κατά κάποιο τρόπο καρπό ε, σοβαρής μελέτης, αλλά θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να αποσαφινιστούν κάποια στοιχεία έτσι ώστε να καταστεί σαφές εάν συνέβη κάτι, αν πραγματικά συνέβη και τι συνέβη. Αυτό που λέμε είναι λοιπόν ότι αυτές οι σοβαρές καταγγελίες ε, θα πρέπει να διερευνηθούν. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και για το ευρύτερο ε, πλαίσιο που θέλετε να δώσετε στη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βαν Όρντεν θα δούμε και εμείς πώς μπορούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στην ε, πολιτική, τη διεύθυνση αυτής της πολιτικής και στις δράσεις σε καθάριση ναρκοπαιδεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να έρθει εδώ ο κύριος Ντεκρέμ. Euh, Συνεχίζουμε λοιπόν τι εργασίε μα, αγαπητοί συνάδελφοι. Με χαρά υποδεχόμαστε τον ε, κύριο Πίτερ Ντεκρέμ, Υπουργό Άμυνα του Βελγίου, ο οποίο θα μα μιλήσει για του έξι μήνε ε, τη Βελγική Προεδρία. Διευκρινίζω αυτή ε, εξ αρχή ότι σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ, βάσει τη Νέα συνθήκη τη Λισαβόνας. Η κυρία Άστον ε, είναι η πρόεδρευσα του Συμβουλίου και αρμόδια για αυτά τα θέματα. Αλλά το σύστημα της εκπεριτροπή προεδρίας συνεχίζεται και έχουν υπάρξει κάποιες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα τη άμυνας ε, το προηγούμενο εξάμεινο το δεύτερο εξάμεινο 2006. Είχαμε για πρώτη φορά επίσημο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνα, ε, ένα μοναδικό σχηματισμό χωρί συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών. Είχαμε άτυπη σύνοδο κορυφή το Σεπτέμβρη στη Γάνδη και σε αυτούς τους διάφορους ε, χώρους, στα διάφορα βήματα συζήτησης, ε, έγινε πολλής λόγος για το θέμα των δυνατοτήτων, για το λεγόμενο pooling and sharing, συγκέντρωση και διαμήραση, επιμερισμός. Και είχαμε και τη γερμανο-σουηδική πρωτοβουλία, την αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανών και Γάλλων, θέματα για τα οποία θα θέλαμε να δούμε μαζί σας ποιες επιπτώσεις είχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της άμυνας διότι είχατε την Προεδρία σε μια μεταβατική περίοδο, έξω και αυτό το ατυπικό κάπο σχήμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ουσιαστικά ε, το Δεκέμβριο του 10 άρχισε να λειτουργεί και αν ε, είχε επικυρωθεί η συνθήκη το 9, το Δεκέμβριο του 9, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμη σε περίοδο προσαρμογής, ιδίως στον τομέα της ΕΠΑ, με διάφορους ορισμούς, Κλοντ Φρανς Αρνό, ε, επικεφαλής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ε, Πρέσβη ΚΟΚ, μόνιμος εκπρόσωπος του ΚΟΠΣ που θα έρθει και στην Επιτροπή μας ε, σύντομα. Ορισμός Γενικών Γραμματέων, παρά τη κυρία Άστον, Ποπόφσκι, στην Επιτροπή μας συγκεκριμένα σύντομα και θέλουμε να μας μιλούν και οι υπουργοί, τα μέλη του Συμβουλίου για την αρχιτεκτονική άμυνας και γενικότερα για τα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Άρα έχετε ένα ευρύτατο πεδίο να καλύψετε. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αρνό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές και λοιποί προσκεκλημένοι. Βρίσκομαι εδώ με πολύ μεγάλη χαρά Απάντησα αμέσως ε, θετικά στην πρόσκλησή σου Αρνό να έρθω να μιλήσω σε εσά για τα θέματα τα οποία με απασχόλησαν το τελευταίο εξάμεινο, το εξάμεινο δηλαδή της ε, Βελγικής ε, Προεδρίας που δεν με απασχόλησαν πια τόσο πολύ τα εγχώρια προβλήματα στα οποία επίσης, τα οποία επίσης αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα στη χώρα. Κυρίε και κύριοι, σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, ε, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει τελείως ε, τα πράγματα. Τα γνωρίζετε κι εσείς, ε, η εκπρόσωπός μας η κάθε Άστον είναι πλέον, έχει πλέον τα ενία σε ό,τι αφορά την αμυντική πολιτική και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και το, τη θέση τη Αντιπροέδρου της Επιτροπής. και είχαμε και ένα θέμα η Βελική Προεδρία υπέρ της εκπροσώπου Άστον. Τρεις λοιπόν, ε, τρία καθήκοντα έχει η κυρία Άστον. Θα πρέπει να συνεχίσει λοιπόν να αναπτύσσει ένα νέο όραμα ε, και ένα νέο όμως ε, σύνολο εργαλείο. Η κυρία Άστον χρειάστηκε να χειριστεί ένα τεράστιο αριθμό φακέλων στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς με πολύ λίγα άτομα. Και ευτυχώς για όλες και όλους φαίνεται να έχει περάσει πλέον αυτή η περίοδος εφόσον πλέον έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, την ΕΙΕΔ. Η δημιουργία της ε, υπηρεσίας μονοπόλησε και μέρος των δραστηριοτήτων της κυρίας Άστον κατά το 2010 και αυτό είχε και επιπτώσεις ό,τι αφορά το χρόνο που στη διάθεσή της για την εξωτερική πολιτική και για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης για το Βέλγιο, ιδρυτικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ανήκουστο στο να μην γεμίσει ο χώρος αυτός και να, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να πάνε στις ελληνικές κάλενδες τα ζητήματα της ε, άμενας ή στο ψυγείο γιατί αυτό είχε βέβαια ε, κινδύνους για μας να μην ξαναβγεί από το ψυγείο το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν την ΚΕΠΑ, έχουμε την ΕΠΑ, ε, πολύ σημαντικά και εκτιμένα της νέας συνθήκης και έναν τομέα κατεξοχήν όπου οι προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης είναι ιδιαίτερε και μεγάλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ε, δεν είναι ένας διπλωματικός εταίρος σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να προχωρήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλη μας την ενέργεια να προχωρήσουμε η ΚΕΠΑ και η ΕΠΑ αναπτύχθηκε κυρίες ε, και κύριοι μέσω της πολιτικής συνεργασίας ε. και συμμετείχαν και οι στρατιωτικές μας δομές σε αρχικό στάδιο για την ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας και αρκετά επιτυχημένα. Έχουμε ένα στρατηγικό δόγμα σήμερα, όχι και τόσο εντυπωσιακό βέβαια, αλλά έχουμε συγκροτήσει και τα απαραίτητα μέσα, μηχανισμούς, δομές για να φέρουμε σε πέρα στο στρατηγικό μας όραμα, είμαστε στη διαδικασία τουλάχιστον. Τα πιο απτά αποτελέσματα όμως είναι οι πολλές αποστολές που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα. Μόλις σε γύρισα από το Τζιμπουτί, όπου είδα ε, την ε, ομάδα μας που, χρησιμο... που συμμετέχει σε μια πάρα πολύ χρήσιμη επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιχείρηση Αταλάντη. Παρέχουμε λοιπόν ε, υπηρεσίες ε, σταθεροποίησης και ασφάλειας και αυτό είναι απαραίτητο για να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και να προωθήσουμε τις αξίες μας. Παρά όμως, τα όσα έχουμε πετύχει, κυρίες και κύριοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι απαιτούνται από την Ευρώπη περαιτέρω προσπάθειε για να είναι ένας υπεύθυνος παγκόσμιος εταίρος και αποτελεσματικό εταίρος. Και θα πρέπει να αναγνωριστεί και να είναι σεβαστή η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, μείζον παίκτη στο διεθνέ προσκήνιο. Η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να κάνουμε μια επικοδομητική συμβολή προ το στόχο αυτό. Προβάλαμε λοιπόν ως βασικό στόχο της Προεδρίας μας ε, την ομαλή και πλήρη υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Πιστεύουμε ως Βέλγιο ότι τα νέα χαρακτηριστικά της συνθήκης μπορούν την κοινή πολιτική ασφάλειας ε, και άμυνας να την οδηγήσουν σε ένα πιο άρτιο και σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ας ξεκινήσω λέγοντας κυρίες και κύριοι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας προτείνει, προβλέπει την καλύτερη υλοποίηση της συνολικής προσέγγισης, του λεγόμενου Global Approach. Μια τέτοια προσέγγιση, συνεκτική προσέγγιση, αποτελεί και ιδιομορφία της Ένωσης, γιατί έχουμε όλα τα μέσα και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να βρούμε με συνεκτικότητα. Η βασική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να συνενώσουμε σε ένα ε, τα στοιχεία ή τέλος πάντων σε περισσότερους του ενός μηχανισμούς ώστε αυτή τη συνολική προσέγγιση να την εφαρμόσουμε και στα θέατρα επιχειρήσεων, όπως τα λέμε, με στρατιωτικούς όρους. Ω Υπουργό Άμυνα θεωρώ ότι ακόμη και η διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων σχεδόν πάντοτε ίσως πάντοτε, τουλάχιστον σχεδόν πάντοτε στο άμεσο μέλλον, θα χρειάζεται και στρατιωτικές δυνατότητες ή στρατιωτική υποστήριξη. Αυτό δεν θα αλλάξει βέβαια τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα, τον πολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη σήμερα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον επιχειρησιακό χαρακτήρα, στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων για, την, ε, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιχειρήσεων. Αυτή η συνολική προσέγγιση λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τομέα και εντό λογικού χρονοδιαγράμματος. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποδέσμη ε, της ε, προσέγγισης αυτής η λεγόμενη πολιτικοστρατιωτική προσέγγιση που θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο είναι η μοναδική πρόταση που έχει να πλασάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να αναπτύξουμε με αξιόπιστο τρόπο αυτές τις μη στρατιωτικέ δυνατότητες, το σχεδιασμό του, την εκτέλεσή τους, ώστε να είμαστε ένας εταίρος επιλογής, ένας ε, απαραίτητος, αναγκαίος εταίρος για τη διαχείριση κρίσεων. Υπάρχει μια μικρή ομάδα συντονισμού η οποία συγκροτείται για τη σταθεροποίηση και ε, την ανοικοδόμηση. Αυτό ε, γίνεται σε επίπεδο ΝΑΤΟ και θα πρέπει και εμείς ως Ένωση να τους δώσουμε τη σωστή απάντηση. Να έχουμε αποτελεσματικέ δυνατότητες που θα μας κάνουν και έναν σεβαστό και χρήσιμο εταίρο και τον είπα. Και αντιστρόφως η ΕΠΑ θα γίνει ένας, ενδιαφ... που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο. Επίσης, έχουμε κάποια εργαλεία, όπως είναι η ρήτρα αμοιβαία συνδρομής ή η ρήτρα αλληλεγγύης. Όλα αυτά είναι στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η ρητρα αλληλεγγυης ολα αυτα ειναι στη συνέχεια της λισαβονας η εσωτερικη και εξωτερική ασφάλεια είναι δύο έννοιες που πλέον ε, αλληλοεπικαλύπτονται θα έλεγα σε κάποιο βαθμό και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια ε, ή την αποκατάσταση ε, καταστροφών. Η παροχή αυτή η αμοιβαία συνδρομή και η αλληλεγγύη είναι σημαντικέ ρήτρε και θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να δώσουμε στι αρχέ αυτέ συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα συνάδει και με το ευρωπαϊκό ε, καθήκον και του ευρωπαϊκού στόχου. Και δεν θα πρέπει να αλληλοεπικαλυφθούμε με τον ΝΑΤΟ. Επίσης, η συνθήκη δίνει και νέες προοπτικές στρατιωτικής συνεργασίας εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΠΕΣΚΟ είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο. Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να δώσει ένα νέο δυναμικό για τα κράτη-μέλη που θέλουν να συνεργάζονται εντός της Ένωσης για να βελτιώσουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες με στόχο την εκτέλεση των πιο απαιτητικών αποστολών. Επί δικής μας Προεδρίας συνεχίσαμε να επεξεργαζόμαστε τις ισπανικές προτάσεις και επενδύσαμε ακόμη περισσότερο στον προβληματισμό και στη σκοπιμότητα να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό τον ε, μηχανισμό, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα να λάβουμε αποφάσεις. Χρειαστούν περαιτέρω προσπάθειες, περισσότερη σκέψη πριν καταλήξουμε σε κοινή συνενός για τον τρόπο με τον ε, οποίο θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολιτική συνένεση. Το κείμενο της συνθήκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει γραφεί πριν από 10 χρόνια περίπου. Το περιβάλλον όμως εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς. Το ΠΕΣΚΟ είναι ένας ε, μηχανισμός, δεν είναι απλά ένα όνομα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εν μέρη έχει ε, επιτευχθεί ο στόχος, όμως το πιο δύσκολο κομμάτι της πορείας μας το έχουμε ακόμη μπροστά μας. Πρέπει να αναπτύξουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τα μέσα τα οικονομικά που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτή τη στιγμή το pooling and sharing είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Αυτό του είδους η συνεργασία σίγουρα προσφέρει δυνατότητες σε λιγότερο ευαίσθητου τομεί, όπω είναι η επιμελητή εκπαίδευση. Ωστόσο, είμαι πεπισμένο ότι αύριο ή ίσω λίγο αργότερα θα δούμε ότι έχουμε ακόμη μεγαλύτερε δυνατότητε και τομεί συνεργασία. Φαίνεται επίση ξεκάθαρο σε μένα ότι δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τη σκέψη μας ή τη φαντασία μας ε, και σε άλλες μορφές συνεργασίας δεν υπάρχει μία μόνο δυνατότητα, υπάρχουν πολλέ. Το περιεχόμενο είναι το σημαντικό και όχι η μορφή. Και πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή ε, προσέγγιση στη συνεργασία. Οποιαδήποτε δηλαδή επιτυχημένη συνταγή θα μπορούσε να επεκταθεί και να επαναληφθεί με άλλου ε, εταίρου. Κυρίε και κύριοι, η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν ε, το εστιακό σημείο της βελγικής ε, πολιτικής στα θέματα άμυνας επί προεδρίας μας. Έχουμε κάποια ε, στοιχεία που διείπαν το εξάμεινό μας. Θέλαμε να είμαστε συνεπείς, αποφασιστικοί, να αντιμετωπίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο τα θέματα που δημιουργούνται από την υλοποίηση συνθήκης της Λισαβόνας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τομέας της άμυνας εν γέννη από τα πρώτα θύματα της ανάγκης ε, εξοικονόμησης ε, των δημόσιων πόρων. Δεν θέλω να ε, χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία αυτό το δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά πρέπει η διεθνής κοινότητα, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτοι από όλους, να ικανοποιηθώ σε αυτό που περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να πάρει τη θέση που έχει ως ένας αποτελεσματικός αξιόπιστος εταίρος. Και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας και των Ευρωπαίων πολιτών με νέα φιλοδοξία, με μειωμένους αμυντικούς προϋπολογισμούς, άρα λιγότερες δυνατότητες και ε, στο πλαίσιο των εθνικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Εγώ, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα, προβληματίστηκα, ίσως και με τολμηρό τρόπο, για το πώς ε, μπορούμε να αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνατότητες ε, πιο, ε, με πιο κοινό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούνται ένα έμβλημα εξοχήν της εθνικής κυριαρχίας των εθνικών κρατών. Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού δεν έχει σε καμία περίπτωση οριμάσει σε πολλά κράτη-μέλη. Η Ευρώπη της άμυνας εντάσσεται παρόλα αυτά σε μια μέρημνα συνεργασίας όλο και στενότερης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, κάνοντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν σταθερό αλλά και αξιόπιστο εταίρο που συμβάλλει στην ασφάλεια, στην ευημερία σε ολόκληρο τον κόσμο και βέβαια πρώτα απ' όλα ε, στη δική μας επικράτεια. Θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα της συνεισφοράς που μπορούμε εμείς να έχουμε στην ιδέα μιας αύξησης των δυνατοτήτων μας με ποιοτική και ποσοτική βελτίωση και αύξηση της συνεργασίας μας έτσι ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές επενδύσεις. Και χρειάζεται επίσης συνεργασία ώστε ναι μεν να εξοικονομήσουμε πόρους αλλά να μην ε, ε, υπάρξουν και αλλοπεκαλύψεις ε, στις διάφορες αγορές εξοπλισμών. Είχαμε τη συμφωνία την αμυντική μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου που δείχνει ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε από κάθε πλευρά είναι η μεγαλύτερη συνεργασία. Η λειτουργικότητα, η βέλτιστη χρήση των στρατιωτικών δυνατοτήτων είναι προφανώς σημαντικά κίνητρα αυτής της πολιτικής ε, εμβληματικής συμφωνίας. Αλλά κατά την άποψή μου δεν χωρεί αμφιβολία για το γεγονός ότι το οικονομικό πλαίσιο το συγκεκριμένο επίσης ε, βοήθησε αυτή την προσέγγιση την τόσο θετική. από την κρίση και από την τρέχουσα κρίση συγκεκριμένα πρέπει εμείς να αντλήσουμε ευκαιρίες. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής, της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι όλο και πιο αισθητέ και στον τομέα της άμυνας και οι επιπτώσεις ε, θα είναι μαζί μας για αρκετό καιρό. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για την άτυπη, για την ανεπίσημη συνάντηση της ΓΑΝΤΗΣ. Κάποιες πτυχές ήταν κάπως ιδιόμορφες δεν ήταν η Λέδη Άστον γιατί ήταν στην κοινοβουλευτική συνέλευση ε, του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ήμουν λοιπόν εγώ αυτός που την αντικατέστησε και έτσι είχα τη δυνατότητα να εφαρμόσω στην πράξη ένα από τα σλόγγαν της Προεδρίας μας με βάση τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Η Βελική Προεδρία στηρίζει την Λέδη Άστον όπως σας είπα και πριν. έχουμε ποιοτικέ εξελίξεις στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Και αυτή ήταν και μία, αυτό ήταν ένα και από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλου που είχε λάβει η χώρα πριν από λίγες ε, ημέρες. Συζήτησαν οι Υπουργοί με τη Λέδη Άστον, το VTC, την ε, προετοιμασία της Υπουργικής ε, Συνάντησης του Δεκεμβρίου και επικεντρώθηκε η συζήτηση στο βασικό θέμα της άτυπης αυτής ε, σύναξης που ήταν οι βελτιωμένες μορφές συνεργασίας, το pooling και sharing των δυνατοτήτων. Κοινές, κοινά ερευνητικά προγράμματα στο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό τομέα. Πώ μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Και αυτό το οποίο προέκυψε από τι συζητήσει είναι η ανάγκη αλλά και η απέτηση ενό νέου πλαισίου, πολιτικού πλαισίου, στο οποίο θα συμμετέχουν όλε οι ήδη φυστάμενε και μελλοντικέ μορφέ συνεργασία. Και ένα κοινό όραμα προσπαθειών. Συμφωνήσαμε όλοι για αυτά τα σημεία και συγκεκριμένα ότι υπάρχει ανάγκη ενός γενικότερου πολιτικού οράματος και κατεύθυνσης και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες Έχουμε τώρα λοιπόν το πλαίσιο Γάνδης. Και ίσω είναι δραματικέ οι εθνικέ επιλογέ που θα πρέπει να γίνουν στον τομέα των δυνατοτήτων. Άρα οι Υπουργοί Άμυνα πρέπει να το έχουν υπόψη και παρόλα αυτά δήλωσαν ξεκάθαρα την πρόθεσή του να εξετάσουν ε, το, τις δυνατότητες αυτές του pooling και sharing. Και αφετηρία τέτοιων σχεδίων θα πρέπει να είναι ότι πρέπει να είναι πρακτικέ και να αυξάνουν την επιχειρησιακή παραγωγή και τα αποχειρησιακά αποτελέσματα. Συζητήσαμε τομεί συνεργασία, στρατιωτική εκπαίδευση, κατάρτιση, διοικητική μέρημνα, μεταφορά, συντήρηση, στοιχεία διοίκηση ελέγχου με το ATC στο Eindhoven ως μοντέλο. Επίσης είχαμε κάποιες ιδέες για τον επιμερισμό ρόλων και καθηκόντων. Αυτό που ισχύει παραδείγματος χάρη στη Βαλτική. Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και σε, άλλους, σε άλλες περιοχές. Η, πολιετής, η πολυκρατική συνεργασία είναι δυνατή, χωρίς όμως να στερηθούν την εθνική κυριαρχία και την ελευθερία δράσης τα κράτη-μέλη. Επίσης, σε ό,τι αφορά ε, μια πολυεθνική μοίρα ελικοπτέρων, ε, και εκεί είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Θα δούμε νέους τομείς συνεργασίας με βάση τις αναλύσεις εθνικών ε, δυνατοτήτων. Ήταν κάτι το υποστηρίχθηκε άλλωστε και γι' αυτό, όπως πρότεινε και ο Γερμανός συνάλφος, συστηματικές αναλύσεις θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι στρατιωτικές μας δυνατότητες. Και είδαμε τρεις άξονες. Πρώτον, ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων των μεμονωμένων κρατών στόχων που θεωρούν ζωτική σημασία και θα πρέπει να παραμείνει στο εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, δυνατότητε συνεργασία, pooling. Τρίτον, στόχοι που μπορεί να ενδιαφέρουν και θα μπορούσαν να ε, επιτευχθούν σε συνεργασία με άλλους εταίρους. Role and task sharing ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα πρέπει να διαδραματίζει έναν σημαντικό και κεντρικό ρόλο στην ανάλυση των δυνατοτήτων και στον εντοπισμό πιθανών τομέων συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και βέβαια το νέο μέσο δεν θα πρέπει αυτό ε, να αποκλειστεί. Μάλλον η δημιουργία νέων μέσων δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εφόσον χρειαστεί στο μέλλον. Το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δεν ήταν το αντικείμενο της συνάντησής μας. Υπουργοί Άμυνα επίση ε, επέστησαν την προσοχή και στον τομέα της αύξησης της αγορά δυνατοτήτων και στην καλύτερη συνεργασία και στην ανάγκη να υπάρχουν λιγότερες στρεβλώσεις και στη δημιουργία ισότιμων όρων. Σε ό,τι αφορά την αγορά εξοπλισμών έγιναν κάποιες προτάσεις και ε, βεβαίως ε, ε, υπενθυμίθηκε εδώ και τα, τα όσα έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό, δημιουργία joint ventures κλπ καθώς επίσης ε, και τα κοινά προγράμματα τα οποία ε, δεν θα στρεβλώνουν τον αναγωνισμό. Όντως ε, διεπίστωσαν οι Υπουργοί ότι το διεθνές ενδιαφέρον βασίζεται στο τοπικό ενδιαφέρον και κυρίως θα πρέπει να έρχεται από, την, από τον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει στην ατζέντα η συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ είναι υποχρεωτική για πάρα πολλά κράτη που είναι μέλη και των διοργανισμών. Πάρα πολλοί υπουργοί υπογράμμισαν ότι η συνεργασία είναι σημαντικότερη από ποτέ. Από κοινού με το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βρει έναν τρόπο για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τη. Εξάλλου πάρα πολλοί υπουργοί θεωρούν ότι είναι σημαντικό να συναντιόνται τα στελέχη του και να ε, δώσουν μια ε, δομή σε αυτές τις συναντήσεις και κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρότεινα στον πρόεδρο της EMC το θέμα αυτό να συζητηθεί με τους εταίρους του του ΝΑΤΟ. Ε, αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Κυρίες και κύριοι, συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι Υπουργοί ε, Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις 9 Δεκεμβρίου του 2010 υπό την Προεδρία της Λέδης Άστον αυτή τη φορά. Συμφώνησαν λοιπόν να επιταχύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, κυρίως δε στον τομέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων. Επίσης ε, συντονίστηκαν βάσει του πλαισίου της ε, Γάνδης ε, όσον αφορά το θέμα της άμυνας σε αυτήν την περίοδο των οικονομικών περιορισμών. Οι συνάδελφοί μου, οι Υπουργοί Άμυνας, συμφώνησαν με το pooling and sharing. Η ΔΕ Γαλλία και η Ηνωμένο Βασίλειο κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησαν ε, την εργασία αυτή μέσω ε, συνεργασίας που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου. Η Σουηδία επίσης ε, έκανε κάποιες νέες προτάσεις όπως έκαναν άλλωστε μέσω επιστολής προς την ύπατη εκπρόσωπο και οι χώρες του Συμφώνου της Βαϊμάρης. Ε, το ε, ΙΑΤΕΣΕ ε, έχει πλέον εγκατασταθεί στην Ολλανδία και αφορά τις τέσσερις υπογράφουσες χώρες. Πρόκειται για μια φιλόδοξη συμφωνία γιατί οι συμμετέχουσες χώρες θα εγκαταλείψουν σε εθνικό επίπεδο τις διαδικασίες ΙΑΤΕΣΕ. Επίσης, ε, στο, ε, στο Βέλγιο ε, υπάρχει η πρόθεση το ναυτικό να είναι πλέον στην υπηρεσία της ΑΠΕΝΕΛ σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική που θέτει θεμέλια για νέα συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Στην άτυπη διάσκεψη του Δεκεμβρίου εγώ ε, ετώνησα ότι όσο περισσότερο, ε, περισσότερη συνεργασία και συντονισμός υπάρχει σε, ευρωπαϊκή, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο και μεγαλύτερο ρόλο θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την ειρήνη και την σταθερότητα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι σημαντική, συνάδει δε και με το κοινό μας μέλλον αλλά και με τους κοινούς μας στόχους. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε αυτήν την συνεργασία με τρόπο ανοιχτό, έτσι ώστε να επιτρέψουμε και σε άλλες χώρες να προσυπογράψουν υπάρχουσες διεργασίες ή πρωτοβουλίες ε, και ε, να αφήσουμε και το περιθώριο για υποβολή νέων πρωτοβουλειών ε, θα γίνει μια έκθεση προς την Λίδια Άστον στα μέσα του τρέχοντος έτους, έτους έτσι ώστε να ε, υπάρξει καλύτερος συντονισμός ε, καθώς επίσης και σωστή κατανομή των πόρων. Κυρίε και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Όπως έχω αναφέρει επανειλημμένα, η πρόοδος ε, στον τομέα των δυνατοτήτων και της άμυνας χρειάζεται νέα όθηση. Η Υπουργή Άμυνας είναι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει έναν ρόλο συντονιστικό σε αυτούς τους τομείς, θα προσφέρει κίνητρα. Θέλουν όλοι να επιθυμούν να συνδράμουν, ε, να συμβάλλουν εργά στη δημιουργία του πλαισίου και επιτρέψτε μου να επαναλάβω τη βούλησή μου και είμαι πεπισμένος ότι η βούληση υπάρχει εκ μέρους όλων των Υπουργών Άμυνας για να στηρίξουμε τις ε, προσπάθειες οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχία της ε, κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Πιέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετικά εξαντλητική ε, παρουσίαση και για αυτή την παρουσίαση της ε, πρωτοβουλίας ε, η Βελική Προεδρία σε υποστήριξη της Λαδής Άστρον που ήταν πραγματικά μια πολύ ενεργητική στήριξη. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν και εγώ όμως να κάνω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Μία πρώτη που αφορά την συνολική προσέγγιση και την στρατηγική εξωτερικής πολιτικής ε, που έχει τη δυνατότητα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, δηλαδή μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική που θα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Την προηγούμενη εβδομάδα ρωτήσαμε την Λέβη Άστον ε, για το Σαχέλ Ε, ε, γιατί θα πρέπει η Υπηρεσία εξωτερική δράση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της απειλής ε, που υπάρχει στην περιοχή Σαχέλ. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την ανάπτυξη, αλλά όχι παραμελώντας την ασφάλεια και την άμυνα. Ε, ρωτώ λοιπόν αυτή η έννοια του επίγοντος χαρακτήρα αυτών των διεργασιών είναι σαφή στο Συμβούλιο. Άλλη ερώτηση για το ΝΑΤΟ. Υπήρξε ε, και η διάσκεψη κορυφή του ΝΑΤΟ στην Λισαβόνα και πολύ μεταξύ ημών απογοητευτήκαμε λίγο όσον αφορά την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Περιμέναμε κάτι καλύτερο μετά από τα πολύ φιλόδοξα αρχικά σχέδια έτσι, εταιρικής ε, σχέσης. Επίσης, το θέμα της Τουρκίας ε, ε, είδαμε ότι δεν προχώρησαν τα πράγματα όπως αρχικά είχε διαφανεί πώς μπορούμε πολιτικά να λύσουμε κάποια προβλήματα ε, και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους πολιτικά ζητήματα ε, ε, να εξουδετερώσουν κατά κάποιο τρόπο τον γενικότερο πολιτικό διάλογο. Τρίτον, αυτό το περίφημο Συμβούλιο Υπουργών, το πρώτο του είδους του, επίσημο Συμβούλιο αποκλειστικά με Υπουργούς ε, Άμυνας. Ε, εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις από ευρωπαϊκής πλευράς. Μετά από αυτή την πρώτη εμπειρία θεωρείς ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή. Εμείς στη δικιά μας ε, έκθεση που κάναμε δηλαδή πέρσι υποστηρίζαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μια διαδικασία συνεχών ε, ε, συμβουλίων Υπουργών Άμυνας, κυρίως όσον αφορά το δυναμικό. Πιστεύεις ότι μετά από αυτό το πρώτο συμβούλιο έχουν αρθεί κάποιες επιφυλάξεις. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Πασκού, θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι η ιδέα αυτή να έρθουμε ένα μήνα μετά ε, το τέλος της ε, Προεδρίας είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Παραδείγματο χάρη, κατά την επόμενη Προεδρία, ένα μήνα μετά το πέρας της Προεδρίας, μπορούμε να καλέσουμε εδώ τον Υπουργό Άμυνα ε, και αυτό να γίνει ένα είδος πεπατημένης, διότι Τότε πια, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η Προεδρία, θα έχει ο υπουργό μια ολοκληρωμένη εικόνα. Έχετε δίκιο λοιπόν κύριε Υπουργέ που είπατε ότι η συνθήκη αυτή ε, είναι πλέον ετών και είναι αρκετά παλαιά. Όμως για αντικειμενικούς λόγους ε, τέθη σε ισχύ μεσούσης της κρίσης. Τι θα γινόταν αν είχε τεθεί σε ισχύ η συνθήκη πριν ξεσπάσει η κρίση. Πάντως τα πράγματα δυστυχώς ε, εξελίχθηκαν όπως σας είπα. Αυτομάτως λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη πόρων και θέλω να πω ότι ανταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές είναι τα τα κράτη της. Όμως, όπως είπατε και εσείς, το μειονέκτημα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα, γιατί με την περίφημη τακτική pooling and sharing, συγκεντρώνουμε σε μια κοινή δεξαμενή και από εκεί μοιράζουμε, ας πούμε με την ε, Γαλλο ε, Βρετανική Συμφωνία υπάρχει είδος, ήδη αυτή η διαδικασία και αν υπάρξει και στο μέλλον θα μας αναγκάσει να αναζητήσουμε μια κοινή διάσταση των θεμάτων κοινού στόχους, κοινά οράματα για ε, πολιτικές και άλλες κρίσεις. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η αξία αυτού του συγκεντρώνω και μοιράζομαι. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε δύο άλλα θέματα. Από ό,τι θυμάμαι στο πλαίσιο της Γάνδης ε, υπάρχει μια πολύ καλή ιδέα ότι ήδη τώρα πρέπει να υπάρχει συντονισμός περικοπών. Δηλαδή υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες είναι διδεθειμένες ε, να προβούν σε περικοπές αμυντικών προβλησμών, λόγω της κρίσης βέβαια. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει κανείς ε, να παρακολουθεί αυτές τις περικοπές γιατί αλλιώς ε, θα καταλήξουμε με χώρες οι οποίες είναι πιο κάτω από το αναμενόμενο επίπεδο ε, κυρίως σε περιπτώσεις και περίοδους κρίσης. Παραδείγματο χάρη, Βουλγαρία, Ρουμανία, αν αυτέ περιέκοπαν δραστικά του προπολογισμού του, τότε αν αυτέ είχαν πρόβλημα θα έπρεπε να επέμβουν οι άλλε χώρε για να λύσουν τα προβλήματά του. Και δεν ξέρω ε, κατά πόσον αυτό είναι αποδεκτό για εκείνου ε, που ε, πιέζονται όλο και περισσότερο. Αν ακολουθήσουμε αυτή λοιπόν την τακτική, ενδεχομένως θα δημιουργηθεί ανισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καταλήξει σε πρόβλημα. Η συνεργασία βεβαίως και στηρίζεται και λόγω της κρίσης. Παράλληλα όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό αντιφάσκει με τον ευρύτερο στόχο που είναι να έχουμε μια ε, κοινή ενιαία αγορά άμυνας. Αυτά λοιπόν που προγραμματίζουμε θα πρέπει, αυτά που προγραμματίζουν όλες οι χώρες δεν θα πρέπει να καταστρέφονται από το ότι δύο-τρεις χώρες αποφασίζουν να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, να καθορίσουν τους δικούς τους όρους, που όμως ίσως να μην είναι αποδεκτοί από όσους βρίσκονται πιο πίσω. Αυτή την ερώτηση είχα να κάνω. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση κύριε Υπουργέ όσον αφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Νομίζω ότι το ευάλωτο σημείο μας ε, είναι το ότι δεν έχουμε κοινή άποψη για την ασφάλεια, άρα δεν μπορεί να υπάρχει κοινή πολιτική για την ασφάλεια. Ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πράξεις δάσης συνεργασίας μεταξύ χωρών, κυρίως μεταξύ χωρών που έχουν σημαντικές στρατιωτικές ικανότητες. Όμως δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ χωρών οι οποίες ε, δεν έχουν ε, το ελάχιστο επίπεδο ε. τι γίνεται όμως, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική όσον αφορά την στρατιωτική ικανότητα κατανοώ τις δυσκολίες, αλλά ε, ξέρω ότι για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε ε, τις, και να αντισταθμίσουμε ε, την, τον αντίκτυπο της κρίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιστοποιήσουμε την χρήση αυτής της υπηρεσίας. Ο κύριος Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ομιλία σας. Νομίζω ότι αυτή η Βελγική Προεδρία σε αυτόν τον τομέα της πολιτικής ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και δημιουργική. Είχαμε πραγματικά ε, μια τεράστια προσφορά κινήτρων και απόψεων από τα κρατη και βεβαίως ε, λόγω της οικονομικής κατάστασης ε, ήταν απαραίτητο να επιδείξετε ρεαλισμό. Πάντως ε, σε πάρα πολλούς τομείς ε, συμβαίνει το εξή ότι λόγω του ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι υπάρχει και μεγαλύτερη προθυμία συνεργασίας. Έχω λοιπόν μια ερώτηση. Καταρχήν όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είπατε ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει λάβει την εντολή να προβεί σε ανάλυση. Σε ποιους τομείς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία. Και είπατε επίσης ποιες χώρες ε, ήδη συνέπτυξαν ε, μορφές συνεργασίας. Αναφέρατε τη Μεγάλη Βρετανία και γνωρίζουμε ότι Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνησή της ε, σκέπτεται του χρόνου ίσως να αποσυρθεί από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Διαφώνησαν με αύξηση του προπολισμού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, μικρή ε, υπηρεσία για του χρόνου. Εσείς όσον αφορά αυτή την υπηρεσία άμυνας, τι πιστεύετε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση γιατί νομίζω ότι θα ήταν λυπηρό η υπηρεσία, η Μεγάλη Βρετανία να αποσυρθεί από την υπηρεσία άμυνας. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω το εξής. Όσον αφορά τη συνεργασία, ε, πράγματι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Μήπως ε, μπορείτε να μας πείτε Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, γιατί αφενός ε, οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε ο ρεαλισμός. Αναφέρατε το European Air Transport Command, αυτό είναι ένα παράδειγμα, και τα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Αλλά ερωτώ, όσον αφορά την μόνιμη μορφή συνεργασίας, ε, πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Και ένα ερώτημα που αφορά σε θέματα προσωπικού. Έχουμε τώρα την ε, νέα διευθύντρια της Υπηρεσίας ε, Άμυνας ε, και μήπως υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ποιος θα καλύψει θέση. Merci, euh, précise qu'il euh, euh, rédige notre rapport CD sur la mise en œuvre. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να αναφερθούμε και στα όσα αναφέρονται στη Λισαβόνα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αλλά και για την ε, πολύ θετική εργασία την οποία ε, έχετε ε, αναπτύξει ως προεδρεύουσα χώρα το προηγούμενο εξάμεινο όσον αφορά την ΚΕΠΑ και την ΕΑ. Ακριβώς στην ίδια γραμμή της αντικειμενικής προσέγγισης που όμως θα βρίσκεται, θα εντάσσεται σε ευρωπαϊκή τροχιά και βεβαίως κατά αυτήν την έννοια ε, είχαμε μία πρώτη πολύ θετική έκβαση της ε, Γάνδης. Ε, παραμένει, παραμένουν βεβαίως πέρα από την προσωπική σας δέσμευση και τη δέσμευση του Βελγίου παραμένει μία τάση ε, περιθωριοποίησης, μία τάση λίγο ολιστηρή όσον αφορά την πολιτική άμυνας και της ε, διαδικασίας ε, προς μια ευρωπαϊκή μια ευρωπαϊκή ε, εξωτερική πολιτική άμυνας και βλέποντας και τις διαδικασίες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια ολίσθηση. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όλους αυτούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο. tre domande sul bilancio del lavoro svolto e anche su sulle indicazioni successivi. Eh, Per quanto riguarda la questione appunto del quadro di Gandhi στα πλαίσια της διαδικασίας της Γάνδης, βεβαίως αναμφίβολα υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό θέμα. Δεν κατάλαβα όμως πολύ καλά τι επιπλέον ε, έδουσαν ε, αυτές ε, οι συμφωνίες των χωρών της Βαϊμάρης, συνεργασίας Γερμανίας, Σουηδίας, πέρα από μια γραφειοκρατική προσέγγιση ας πούμε. Και εγώ θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω την σημασία του να περάσουμε από τα λόγια, από τα paper, χαρτιά, έγγραφα και ξανά χαρτιά, από τα λόγια λοιπόν και από τα γραμμένα στις πράξεις γιατί ξέρετε σε έξι μήνες θα έχουμε ένα νέο κατάλογο, ε, θα έχουμε καταλόγους επί καταλόγων, λίστες επί λιστών και από εκεί και πέρα καμία δουλειά συγκεκριμένη. Η δεύτερη, το δεύτερο ζήτημα αφορά τον συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες δομές οι οποίες ασχολούνται με την αντιμετώπιση των κρίσεων καθώς επίσης ε, και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία παραμένουν ακόμα εκρεμή. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει έτσι ώστε να ενισχύσουμε την, ε, ε, να ενισχύσουμε τις, ε, τα στρατιωτικά μέσα. Το ζητάει το Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να καλυφθεί η ε, διάσταση ανάμεσα στην ε, μη στρατιωτική λογική των στρατιωτικών διεργασιών και ε, την συνεργασία κατά κάποιο τρόπο, το κλείσιμο της ψαλίδας με την στρατιωτική αντιμετώπιση. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταφ. Um, <coughs> President, um,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 Χαίρομαι πάρα πολύ για τη Συμφωνία Αγγλογαλλικής ε, Συνεργασίας ε, που όπως είπατε είναι μια συμφωνία πολιτική αλλά και πρακτική και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως ε, είναι ξαλού και μια συνθήκη, ας το πούμε αυτό, που είναι εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία η οποία επίτηδες μάλιστα βγαίνει από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό, το κρίνετε ως πρόκληση, πιστεύετε ότι κατά κάποιον τρόπο η συμφωνία αυτή υπονομεύει τη λογική που διέπει τη συμφωνία της Λισαβόνας και ερωτώ ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι υπόλοιποι Υπουργοί Άμυνας των 25 κρατών σε αυτή την ε, γαλλοβρετανική συνεργασία. Στην πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι Υπουργοί Άμυνας της ε, Γαλλίας ε, και της Γερμανίας να παρουσιάσουν αυτό το τετελεσμένο γεγονός. Όσον αφορά το στρατηγικό, τη στρατηγική διάσταση, για πρώτη φορά μοιάζει να υπάρχει μια στρατιωτική στρατηγική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα υπάρχει εμπλοκή ε, της τουρκοκυπριακής διένεξης. Πρόκειται για ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, όπως είπε και ο πρόεδρος. ένα τεράστιο κόλλημα που παρεμποδίζει τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εγώ όμως, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ, σύντομα πρόκειται να επιληθεί ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί και υπάρχει βέβαια και το ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα του Ιράν. το όλο θέμα φεύγει από τα ακαδημαϊκά σεμινάρια. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν ορισμένες συζητήσεις για θέματα άμυνας ε, ανάμεσα στα κράτη. Μοιάζουν με ακαδημαϊκά σεμινάρια οι συζητήσεις αυτές και το όλο θέμα μπαίνει στον, στο πεδίο της πρακτικής πολιτικής. Εσείς πώς το βλέπετε, πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να έχουμε ενωμένη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ απέναντι στην πρόδειλη αποφασιστικότητα του Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη, το σχεδιασμό πυρηνικής βόμβας. Ο κ. Πιτικόφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ επίσης κύριε Υπουργέ για τις εκτενείς ε, παρατηρήσεις σας και έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη έχει σχέση με αυτά που είπαν οι κύριοι Γκάλα και Νταφ. Και εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει ποια προβλήματα προκύπτουν ή εκρεμούν ακόμα και πρέπει να επιληθούν όσον αφορά αυτή τη δομή της μόνιμης συνεργασίας. Εσείς είπατε στα αγγλικά ότι αυτό που χρειάζεται ακόμα είναι more new thinking, κάποιες ρηξικέλευτες δηλαδή απόψεις. Και αυτό με ενδιαφέρει κατά πόσον αυτό σχετίζεται με αυτό που είπε ο κύριος Νταφ. Δηλαδή η ιδέα της μόνιμης δομημένης συνεργασίας, εξορισμού, είναι ευρύτερη, συμπεριληπτική, αν μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ενώ η άποψη της Γαλλίας και της Βρετανίας είναι αποκλειστική, αποκλείει πράγματα, διάσταση θεμάτων. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα συνδυάσει όλα αυτά πολύ συμπατικά και φιλικά όπως το κάνατε εσείς με ιδιαίτερα ε, διπλωματικό τρόπο. Ε, το κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε και στο μέλλον. Αλλά αν μιλήσουμε επί της ουσίας, πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε ώστε τέτοιου είδους ε, τάσεις αποκλεισμού να μην παρεμποδίζουν μια ανοιχτή διαδικασία συμπερίληψης. Και αυτό που με ενδιαφέρει επίση είναι και το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο εντάσσεται η EDA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και κάνει τις αναλύσεις της που αφορούν στο ε, δυναμικό περαιτέρω συνεργασίας. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο, εγώ πιστεύω στις Γερμανο ε, σουηδικέ προτάσει σχετικά με το pooling και sharing και εκεί ξεκολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ας πάρουμε ε, το θέμα της Γερμανίας χάρη. Εκεί το ε, Κοινοβούλιο έχει επιφυλάξει όσον αφορά την ανάπτυξη γερμανικών δυνάμεων. Ε, ίσως τα προβλήματα να είναι μικρότερα στο pooling, αλλά όχι τόσο στο sharing. Και με ενδιαφέρει λοιπόν κατά πόσον τέτοιου θέματα συζητήθηκαν. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Πολύ σωστά επισημάνατε αυτή την ε, κινητήρια δύναμη που τελικά συνεπάγεται ο περιορισμός πόρων. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον οι Υπουργοί Άμυνας θα κάνουν ένα βήμα παραπάνω, κατά πόσον θα εκμεταλλευτούν αυτή την κινητήρια δύναμη έτσι ώστε να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο στη συνεργασία με τρίτους. Ας πούμε το ΝΑΤΟ αποφάσισε στη Λισαβόνα ότι πρόκειται να αναπτύξει περαιτέρω την αστική διάσταση των προγραμμάτων του. Και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει έγκαιρα με το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε στην περίπτωση που το ΝΑΤΟ να λάβει δικές πρωτοβουλίες να μην υπάρξει επικάλυψη. Ή άλλο παράδειγμα, Αταλάντα. Αν ας πούμε σκεφτούμε την εθνικότητα των σκαφών που προστατεύονται από την πειρατεία. Θα μπορούσε κανείς να καταλήξει το συμπέρασμα ότι η Κίνα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη εισφορά. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό που συνεισφέρουμε εμείς ε, δεν βρίσκεται σε αναλογία με αυτό που ε, συνεισφέρει η Κίνα αν λάβει κανείς υπόψη του τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται. Αυτό σας ενδιαφέρει ή και στην περίπτωση της Ρωσίας η συνεργασία με τη Ρωσία. Εκεί σε αυτή τη συνεργασία μπορεί να προκύψει κάποια εξοικονόμηση πόρων. Το τελευταίο μου ερώτημα αφορά το Σουδάν. Υπήρξαν άραγε σκέψεις να ασχοληθείτε με το Σουδάν εφόσον κάτι τέτοιο ε, κρυθεί απαραίτητο. Ελπίζουμε όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει εξεταστεί αυτή η περίπτωση. Η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω κατ' ουσίαν τις ερωτήσεις του κυρίου Πιουτιχόφα. Όσον αφορά το θέμα του κόστους, ε, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτή την ένταση που προκύπτει ανάμεσα στην αναγκαιότητα εξοικονόμησης πόρων αφενός και αφετέρου στις ε, υποχρεώσεις ε, αγοράς ε, εξοπλισμών και παρεμφερή. Τα προγράμματα εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τελευταίο καιρό ήταν πολύ συγκρατημένα. Υπάρχει πράγματι μία τάση εξοικονόμησης ενταπανών, αλλά τον τελευταίο καιρό υπάρχει το Α400M και το ελικόπτερο Τίγρης. Ε, ακούγονται αυτά. Και γι' αυτό ερωτώ, εσείς κατά τη διάρκεια της δικής σας της ε, θητείας, τι κάνατε για να αντιμετωπίσετε αυτή την τάση που διαφαίνεται πλέον καθαρά. Ε, το επόμενο ερώτημά μου αφορά την ρήτρα αλληλεγγύης. Αναφερθήκατε κι εσείς σε αυτήν και κατά την άποψή μου ε, πολλοί αποκρύπτουν, αγνοούν αυτή την ρήτρα. Και εσείς μιλήσατε για ε, προβλήματα διαχωρισμού είπατε ότι πρέπει να διαχωρίζεται η εξωτερική ασφάλεια από την εσωτερική ασφάλεια που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, σε τελική ανάλυση, τι ακριβώς γίνεται με θέματα ασφάλειας στο πλαίσιο της ε, ρήτρας ασφαλείας. Ε, σε αυτές ε, τις περιπτώσεις ασφάλειας εμπίπτουν εκεί οι διαμαρτυρίες ή, ας το πω αλλιώς, αν σε κάποια, κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κατάσταση όπως αυτή που προέκυψε στην ε, την Ισία. Θα παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει το πρόβλημα, να προστατεύσει τους ε, ανθρώπους. Ή στο θέμα της ελευθερίας τύπου, η ρήτρα αυτή ασφαλείας, τι ακριβώς προβλέπει, τι θα μπορούσε να γίνει. Ερωτώ λοιπόν πώς ακριβώς προκύπτει αυτός ο διαχωρισμός και πώς ορίζονται οι ε, καταστάσεις, οι συνθήκες ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν ό,τι είχα να πω έχει υποθεί. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την ε, παρουσία του και για την ομιλία του που ακούγοντάς την ένιωθα πραγματικά ευτυχής και σε ταύτιση με αυτή την τόσο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση. Και ήθελα να πιστεύω ότι είναι και όλα αλήθεια. Δεν εννοώ ότι είπατε ψέματα, κύριε Υπουργέ. Απλά από την πρακτική η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι για συγκεκριμένες χώρες και για μία μειοψηφία βουλευτών, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται όμω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα τη ασφάλεια και τη άμυνα εξακολουθεί να είναι το όριο, το ανυπέρβλητο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σε ό,τι αφορά την κοινοτικοποίηση των πολιτικών. Και δυστυχώ το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Με τέτοια συχνότητα που δεν είναι δυνατόν ε, πλέον να το επιλύσουμε. Δεν το έχουμε επιλύσει ακόμη. Είδαμε το πλαίσιο της Γάνδης, το Συμβούλιο, τι είπα, αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος ή άλλοι συνάδελφοι, Γκουαλτιέρη, Νταφ, θα πω και εγώ με άλλα λόγια το ίδιο, ότι δηλαδή εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απόφαση από πλευρά Συμβουλίου ή είπα της εκπροσώπου, αλλά ούτε και από την πλευρά των αδελφών οργανισμών όπως είναι η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να δείχνει ότι έχουμε υπερβεί αυτό το όριο που φαίνεται ότι είναι ανυπέρβλητο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, πρέπει να υπάρχει επιμερισμός ε, των μέσων της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ακόμη και σήμερα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τους υπουργούς, ιδιαίτερα εξωτερικών αλλά και άμυνας, να ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες, σε περιοχές τρίτων χωρών του κόσμου και μιλούν για τη δική τους χώρα, εξ ονόματος της χώρας τους, όχι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως είναι κοινοτοπία να το ξαναπώ, αλλά δεν μιλάνε με μια κοινή φωνή, δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική, δεν υπάρχει ένα κοινό όραμα για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Έχετε γύρω στα 10 λεπτά, δεν είναι πολύ ο χρόνος για να απαντήσετε. Φαντάζομαι όμως ότι επειδή πολλά θέματα είναι αλληλοσυνδεόμενα, μπορείτε να είστε συνθετικός. Πολύ λίγες ερωτήσεις, πολύ λίγος χρόνος, δυστυχώς λέει ο Υπουργός. Λίγες απαντήσεις ε, σύντομες μάλλον, οι οποίες όμως ελπίζω ότι θα απαντήσουν ικανοποιητικά στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν. Πρώτα απ' όλα, θα δω λίγο όλες τις ερωτήσεις ε, που ετέθησαν. Γιατί πολλές συγκλίνουν από τις ερωτήσεις. Πρώτον, η ε, συνολική προσέγγιση ε, νομίζω ότι ε, αποτελεί μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση που αφορά όλα τα ζητήματα. Ας πούμε το θέμα το οποίο εθέσατε για την περιοχή του Σάχελ. Ήμουνα στο Μαρόκο την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί στο Μαρακές ε, ζήτησα να υπάρχει συνολική προσέγγιση του θέματος έτσι ώστε να είναι λειτουργική. Συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η συνεργασία ε, είναι απαραίτητη ε, και αφορά την ασφάλεια των στρατιωτών μας πρώτα απ' όλα. Εγώ είμαι εδώ και σαν Υπουργός εξωτε... Ε, συγγνώμη, Άμυνας, ο οποίος διπλασίασε το δυναμικό σε άνδρες στο εξωτερικό. Η συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη έτσι ώστε ε, να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των στρατιωτικών μας ε, και για να ε, παραφράσω τον Γουλιέλμο τον Σιωπηλό μπορώ να πω ότι δεν, δεν είναι απαραίτητο απλώς να έχουμε μια βροντερή προσέγγιση, πρέπει να έχουμε μια καλή προσέγγιση. Συμβούλιο Άμυνας. Πολλές ερωτήσεις για το Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ δεν διάβασα πουθενά οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε έντυπο εφημερίδα, ε, δεν άκουσα κανέναν ε, αρχηγό πολιτικής ομάδας, ε, οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας στο Κοινοβούλιο, που να μην λέει ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος η ανάπτυξη της, της άμυνας. Είναι επομένως ισχυρός ακρογωνιαίος λίθος για για οποιοδήποτε ευρωπαϊκή ε, πολιτική. Επομένως η συνεδρίαση αυτή, το συμβούλιο αυτό ε, ήταν ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Κοιτάξτε, δεν μετακίνησε, δεν τάραξε με οποιοδήποτε λόγο την ορθοδοξία των απόψεων, άλλωστε δεν είχε τέτοια δογματική προσέγγιση ή φιλοδοξία, δεν ξεπεράσαμε σκαμμένα, δεν ξεπεράσαμε όρια όμως ήταν μια καλή αρχή. Πιστεύω ακράδαντα λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί ακριβώς μέσω τέτοιων ε, συνεδριάσεων ε, θα ε, καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτήν την κοινή οπτική και κοινή προσέγγιση. Όσον αφορά την ΕΠΑ, από την ε, σύλληψή της αλλά και λόγω της ε, άποψης που συμμερίζονται οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι ένα φιλόδοξο εργαλείο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει, πώς να σας το πω, ε, να το δούμε φιλόδοξα. Γιατί μέχρι τώρα δεν καταφέραμε να δούμε πολύ καθαρά περί τίνος πρόκειται και ενδεχομένως δεν υπάρχει μονάχα μία, ένα όραμα, ίσως το όραμα να είναι μολταπλό, ε, συγγνώμη, πολλαπλό. Ε, πρόκειται για μία πολύ σημαντική διαδικασία. Πρέπει να δούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, όλους τους εμπλεκόμενους, ε, έτσι ώστε το όραμα να συνεχιστεί και να ε, διευρυνθεί. Ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ε, υπηρεσία ασφάλειας. Έγινε λόγος ε, και ε, στην προηγούμενη συνάντηση. Η κυρία Αρνό είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επικεφαλής πλέον αυτής της υπηρεσίας, της ΕΝΤΑ. Ε, με τεχνικά θέματα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ασχοληθεί η ΕΝΤΑ. Πέραν αυτού όμως στη Γάνδη ε, σαφώς ε, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να έχει και μια συγκεκριμένη στρατηγική, δηλαδή να ζητήσουμε από την ΕΝΤΑ να έχει περισσότερη ε, φιλοδοξία. Μία τέτοια λοιπόν υπηρεσία πρέπει να έχει, οφείλει αλλά και μπορεί να έχει, γιατί ε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχει μεγαλύτερη ε, ε, φιλοδοξία. Άλλες ερωτήσεις πάντα για τη Γάνδη, για το πλαίσιο της Γάνδης. Qui sont, qui sont donc pour des opérations, euh, υπό την ευρύτερη ε, κάλυψη της Ευρώπης ε, ακούγονται πολλά, όλο και πιο αξιόπιστα και όλο και πιο αποδεκτά όσον αφορά την συνεργασία και όσον αφορά μία κατά κάποιο τρόπο αλληλεξάρτηση η οποία οριμάζει ακόμα περισσότερο ε, τις προτάσεις. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε ε, μια θετική ανταπόκριση σε ένα αίτημα συνεργασίας, τότε διευρύνεται, γίνεται πιο αξιόπιστη αυτή η συνεργασία. Όσον αφορά τον συνάδελφο κύριο Ντάφ. Ξέρετε ότι ήμουν ε, πολύ ευγενή ε, κατά την παρέμβασή μου, ίσως να μην συμφωνείτε όλοι με αυτό που λέω, αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, συνηθίζω ε, το 99% των περιπτώσεων να είμαι ευγενή ε, στι παρεμβάσει μου. Νομίζω λοιπόν Μάλλον, ε, να το πω αλλιώ. Ε, πράγματι, η συμφωνία αυτή ανάμεσα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντική και δεν νομίζω ότι βγαίνει από το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Ε, μιλάμε για δύο χώρε κλειδί τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στο κέντρο αυτή, είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και ό,τι και αν πιστεύει κανεί ή αν επιθυμεί, ε, κανεί δεν είναι ποτέ εκτό της διαδικασίας σίγουρα όχι στα στρατιωτικά θέματα. Νομίζω ότι αύριο θα μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα από ό,τι σήμερα και η συνθήκη αυτή είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έλεγα λοιπόν ότι ε, θα ήταν κρίμα να αντιμετωπίζει κανείς αυτό το βήμα ως ένα βήμα εκτός ε, του πλαισίου στρατιωτικής συνεργασίας. Όσον αφορά στο Ιράν, Νομίζω ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ε, τεράστια πρόκληση, η οποία όμως ε, προσφέρει και ευκαιρίες και προσφέρει και την ε, δυνατότητα κοινή αντίδρασης ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην στατική του ΝΑΤΟ για εμπλωτισμό ουρανίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση Και όσον αφορά τα άλλα θέματα που αναφέρατε, για την Αταλάντα πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη διαδικασία και το ερώτημα που τίθεται είναι ε, για πόσο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται εκεί ε, στο κέρας της Αφρικής. Εγώ αντιμετωπίζω την επιχείρηση ε, στο σύνολό της και νομίζω ότι μέχρι το 2012 θα παραμείνει εν ζωή. Τα κρατη την κρίνουν επιτυχημένη την επιχείρηση αυτή. Κατ' ουσίαν πρόκειται για σταθεροποίηση, για μια επιχείρηση σταθεροποίησης μέσω ε, στρατιωτικής ε, παρουσίας και κάθε φορά που έχουμε την δυνατότητα να συναντήσουμε συναδέλφους σε άλλο πλαίσιο αυτό είναι θετικό, είναι μια ε, επιχείρηση όπου εκεί παραδείγματος χάρη μπορεί κανείς πράγματι να δοκιμάσει το πώς αποφεύγονται οι επικαλύψεις. Νομίζω ότι απάντησα στις ε, περισσότερες ερωτήσεις. Η τελευταία μου απάντηση αφορά στην ερώτηση του συναδέρφου Λέζινγκ. Σε ό,τι αφορά που είναι η συνάδελφο Λέζινγκ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αλληλεγγύη, πολύ σημαντική ρήτρα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη για να επεξεργαστούμε τη ρήτρα αυτή. Κάτι που πρέπει να αποφύγουμε όμως κατά την άποψή μου και ισχύει και για τον ΝΑΤΟ αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θεωρούμε θεός μελλοντική αστυνομία ή αστιφύλακες που θα ε, διαφεντεύουμε στον κόσμο, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επεξεργαστούμε τη ρήτρα αλληλεγγύης και εκεί να καθορίσουμε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, ε, που τη δώσατε τις, τις απαντήσεις σας και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχαμε. Συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασαν πολλοί συνάδελφοι και ο Αντιπρόεδρος Πάσκου μεταξύ αυτών για την χρησιμότητα ανταλλαγών απόψεων και απολογισμών σαν αυτών που μας δώσατε για την Βελική Προεδρία. Και μας άρεσε αυτό που είπατε ότι η Βελγική Προεδρία στηρίζει τη Λέδη Άστον. Είναι ο σωστός, η σωστή φόρμουλα και ελπίζω να σας ξαναδούμε και σύντομα για να δούμε τι γίνεται και στα θέματα της ε, ΚΕΠΑ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ τις εργασίες μας. Την Πέμπτη το πρωί δεν έχουμε συνεδρίαση, άρα την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου θα ξανασυνεδριάσουμε.